colleagues, I like to start the meeting. everybody can stay with Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αρχίσουμε. Σας καλωσορίζω λοιπόν όλους όσοι βρίσκεστε εδώ. Μερικοί από εσάς έχετε ξανάρθετε, ξανάρθει εδώ, οπότε καλώς ήρθατε και πάλι. Έχουμε από 24 χώρες μέλη ευρωβουλευτές, αλλά έχουμε και από τρεις υποψήφιες χώρες, την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και την Τουρκία και έχουμε επίσης και από την Νορβηγία που είναι από τις χώρες ΕΖΕΣ. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε για να συζητήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι πολύ καλή εκπροσώπησή μας εδώ. Έχουμε και εκπροσώπηση της Αυστριακής Προεδρίας, την κυρία Τζουλιάν Μπόγνερ Στράους, που είναι υπουργό στην Ομοσπονδιακή Καγκελερία για Γυναίκες, Οικογένεια και Νεολαία. Και έχουμε και την Επίτροπο Βέρα Γιούροβα, η οποία είναι υπεύθυνη για την δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Έχουμε και το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Έχουμε μαζί μας ε, τον Ρέιν Λόπατκα, που είναι πρόεδρος της ε, Μόνιμης Υποπιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και τον Κρίστιαν Πούχμαν, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου. Περιμένουμε ακόμα και τον πρόεδρο της ΟΚΕ, τον Λούκα Ζαγέ. Έχουμε ε, επίσης την Επιτροπή των Περιφερειών, την κυρία Μπάρμπαρα Ντούντεν, που είναι πρόεδρος ε, της Επιτροπής που ασχολείται με τα θέματα ηθαγένεια, διακυβέρνηση θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις Και περιμένουμε και τους εμπειρογνώμονές μας. Έχουμε, από Έχουμε μάλλον ένα προσκεκλημένο εμπειρογνώμονα που είναι ο Γουακίν Αλμούνια, τον ξέρετε, ήταν παλιά επίτροπος. Και να σας υπενθυμίσω ότι σε αυτό το σύστημα διακοινοβουλευτικής επιτροπής συνεδριάζουμε κάθε χρόνο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Μια φορά το χρόνο κανονικά. Και περί τίνος πρόκειται, θέλουμε να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε μια κοινή ευθύνη απέναντι στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να διαμορφώσουμε το σώμα για το μέλλον Άρα πρέπει να προβληματιστούμε για το μέλλον της Ευρώπης και να αναλάβουμε και τις ευθύνες μας όσον αφορά τη στήριξη των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Εκλογόμαστε με καθολική ψηφοφορία, οπότε εμεί εκπροσωπούμε τους λαούς μας και η φωνή τους πρέπει να εισακούεται κάθε φορά που παίρνουμε αποφάσεις. Και εσείς έχετε την υποχρέωση να ελέγχετε τις κυβερνήσεις σας, την εκτελεστική εξουσία δηλαδή στις χώρες σας, αλλά και εδώ εμείς ελέγχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό για όλους μας και πρέπει να είμαστε σε θέση να δείξουμε στους πολίτες ότι εμείς που εκλεγόμαστε από αυτούς μπορούμε και επηρεάζουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φέτος λοιπόν βρισκόμαστε εδώ για να ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ μας όσον αφορά την κατάσταση πραγμάτων και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως γνωρίζετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε τρεις τάσεις συζήτησης ανεξάρτητες. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη Λευκή Βίβλο και ό,τι ακολούθησε όσον αφορά την κατάσταση πραγμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ήταν η ομιλία του Προέδρου της Jean-Claude Juncker. Άρα έχουμε το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προβληματισμό αυτό. Στη συνέχεια έχουμε τη συζήτηση και κάποιες αποφάσεις που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο, και έχουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου και εδώ συζητούμε και προβληματιζόμαστε για την μορφή που θα έχει η μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίσαμε το 2017 με την έκθεσή μας και τώρα δουλεύουμε πάνω σε μία έκθεση που θα είναι η κληρονομιά που θα αφήσει η κοινοβουλευτική μας αυτή η Επιτροπή για το μέλλον. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη και τα τρέχοντα γεγονότα. Η Προεδρία της Επιτροπής με την κατάσταση πραγμάτων στην Ένωση, ο Ζαν Κλώτο Γιούνκερ είπε ότι θα έρθει με προτάσεις προκειμένου να επεκταθεί κατά κάποιο τρόπο η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε περισσότερους τομείς πολιτικής. Ε, μιλήσαμε επίσης και μίλησε και εκείνος τότε για τη διαφάνεια, όχι μόνο εδώ, αλλά και στο Συμβούλιο. Σε συνεργασία μάλιστα με τον Ombudsman, με την Ombudsman. Και επίσης θέλουμε να αγωνιστούμε και για κάτι που για σας μπορεί να είναι καθημερινότητα, αλλά είναι οι ερευνητικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δυστυχώς δεν έχουμε πείσει τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα ότι αυτό το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί σε αυτή τη θητεία. Εδώ θα ακούσετε από τους συναδέρφους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις εκθέσεις μας. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τη συζήτηση αυτή την κάνουμε μαζί σας, αφού προηγουμένως βέβαια έχει γίνει πολύ προκαταρτική δουλειά. Χωρίς λοιπόν άλλη καθυστέρηση και πριν δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας, θέλω να σας ενημερώσω για κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες. Κάποιοι από εσά μπορεί ήδη να τα γνωρίζετε, αλλά βλέπετε έχετε κάτι χαρτάκια μπροστά σας, στα έδρανά σας, που πρέπει να τα συμπληρώσετε αν θέλετε χρόνο ομιλίας να πάρετε το λόγο δηλαδή εδώ στη συζήτηση. Θα τα συγκεντρώσουν ε, κλητήρες, θα φτάσουν εδώ σε εμά και έτσι ανάλογα με το πόσοι θα έχουν ζητήσει το λόγο θα φροντίσουμε και για την αντίστοιχη κατανομή του χρόνου ώστε να μιλήσουν και βουλευτές από τα Εθνικά Κοινοβούλια και ευρωβουλευτές. Ο πρώτος που θα πάρει το λόγο εκ μέρους της Προεδρίας είναι η Υπουργός Τζουλιάν Μπόκνερ Στράους. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much. Σας, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Χίμπνερ, Πρόεδρε της Επιτροπής ΑΦΚΟ, κυρία Επίτροπε Γιούροβα, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου τιμή να εκπροσωπώ εδώ την ε, Αυστριακή Προεδρία για να συζητήσουμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι αυτές οι συναντήσεις ανάμεσα στις Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις Επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων είναι πάρα πολύ μεγάλης σημασίας για να ενισχυθεί ο διάλογος και να συζητηθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η Αυστρία επικροτεί τον ενεργό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη συμβολή του στην συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι συζητήσεις υψηλού επίπεδου όπου καλούνται οι κυβερνήσεις ε, των κρατών μελών είναι πολύ σημαντικοί διότι ε, το, η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Ε, ζούμε σε εποχή με αναταράξεις και χρωστάμε στους πολίτες μας μια ειλικρινή συζήτηση σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα για να προστατεύσουμε τα επιτεύγματα μιας ενωμένης και ειρηνικής Ευρώπης. Θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία σήμερα για να σας παρουσιάσω σύντομα τις απόψεις της Αυστριακής Προεδρίας για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στην ε, συνέχεια της επιτυχίας της Ευρώπης. Το σύνθημά μας είναι μια Ευρώπη που προστατεύει και στόχο έχει ε, να ε, διασφαλίσει την ασφάλεια, να λύσουμε την πρόκληση της μετανάστευσης και να έχουμε σταθερότητα στις γειτονικές χώρες. Αυτές είναι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών μας. Όσον αφορά την ασφάλεια και τη μετανάστευση, την πρώτη μας προτεραιότητα, εργαζόμαστε σκληρά και με επιμονή για να ε, έχουμε επιτυχία. Οι συζητήσεις ε, στο Σάλσπουργκ έδειξαν ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής ε, σχετικά με τις επιστροφές και την προστασία των συνόρων θα πρέπει να εξεταστούν ε, και να θεωρηθούν προτεραιότητα. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η βούλησή μας να συνεργαστούμε πιο στενά με τις χώρες Αφρικής. Την επόμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξετάσει αυτά τα θέματα και ο καγκελάριος Κούρτς θα εξετάσει το κοινό σύστημα ασύλου και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα διάφορα στοιχεία του συστήματος αυτού. Επίσης, η ψηφιακή ενιαία αγορά ε, είναι πολλά υποσχόμενο εγχείρημα. Ξέρουμε ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες και τα ψηφιακά επιχειρηματικά πρότυπα ε, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Πρέπει να δημιουργήσουμε το σωστό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, για να μπορούν να ευημερίσουν και να αναπτυχθούν ασφαλής ένωση μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον είναι ασφαλής όλη η περιφέρεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε ψηλά στο πολιτικό μας θεματολόγιο την προσχώρηση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Θα πρέπει αυτό να γίνει με σαφή κριτήρια που να έχουν να κάνουν με τις επιδόσεις της κάθε χώρας και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να έχουμε απτή πρόοδο. Το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν θα ολοκληρωθεί εάν δεν ε, ενσωματωθεί πλήρως όλη αυτή η περιοχή. Επίσης, έχουμε εντατικές συζητήσεις σχετικά με τις προτάσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στηρίζουμε τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, επιτευχθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσης, πρέπει να ε, ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και να κερδίσουμε και την εμπιστοσύνη των νέων. Το σενάριο 4 θεωρήθηκε ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασχολείται με τα μεγάλα προβλήματα όπου χρειάζονται μεγάλες λύσεις. Οι περισσότεροι όμως δεν θέλουμε μια Ευρώπη που να εμπλέκεται σε κάθε μικρό πρόβλημα όπου είναι καλύτερο να αποφασίζουν οι τοπικές αρχές και οι περιφέρειες. Γι' αυτό πρέπει να ενισχυθεί η αρχή της επικουρικότητας. Επικροτούμε τα αποτελέσματα της ειδική ομάδας εργασίας για την επικουρικότητα και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις στις 15 και 16 Νοεμβρίου στο Πρέκενς. Η ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών είναι ένα προσβάσιμο εργαλείο για τους πολίτες ε, ώστε να μπορέσουν να επηρεάσουν το θεματολόγιο. Όπως και άλλα κράτη-μέλη, έχουμε διαβουλεύσεις με τους πολίτες μας. Οι διαβουλεύσεις αυτές ε, θα μας δώσουν πολύτιμα στοιχεία για τη συνέχιση της συζήτησης σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τα θέματα νεολαία Πρέπει να θυμόμαστε ότι η νεολαία είναι και το μέλλον της Ευρώπης. Δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα τις εργασίες μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή θα οικοδομηθεί από τη σημερινή νεολαία. Επίσης θα ήθελα να τονίσω κάτι εξίσου σημαντικό. Οι νέοι είναι και το σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η απτή επιτυχία ε, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ε, καταδεικνύεται περισσότερο από πουθενά αλλού από το πρόγραμμα Εράσμους. Γνωρίζουμε ότι στο δημοψήφισμα για το Brexit οι νέοι ψήφισαν ε, κατά μεγάλη πλειοψηφία το να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη δική μου χώρα πάνω από το 80% των νέων Αυστριακών νιώθουν ότι είναι Ευρωπαίοι. Ταυτόχρονα θα πρέπει να φροντίσουμε να ακουστεί η φωνή των νέων και να ληφθεί υπόψη. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Η άτυπη συνάντηση στη Βιέννη αρχές Σεπτεμβρίου με υπουργού νεότητας πρώτη από το 2006 συνδυάστηκε με την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νεολαίας. Ε, εκπρόσωποι των νέων μπόρεσαν να συναντηθούν με τους υπουργούς και να ε, συζητήσουν τα θέματα που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Κυρίες και κύριοι, ε, τώρα ξεκινάει η κρίσιμη συζήτηση για τις εκλογές του Μαΐου του 2019 και πρέπει να γνωρίζουμε τις βασικές προκλήσεις και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να τα αντιμετωπίσουμε. Προσβλέπω στην ε, παρουσίαση του κυρίου Αντώντο σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Προχωράμε στην κυρία Επίτροπο, την κυρία Γιούροπα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, με τα χαρά σας παρευρίσκομαι εδώ σήμερα και είναι προνόμιο για μένα να μιλήσω για το θέμα αυτό. Όταν το πρωτοδιάβασα, uh, αισθάνθηκα έτσι μια ανησυχία. Το μέλλον της Ευρώπης, ποιος μπορεί να το ψυχανεμιστεί. Λοιπόν, άρχισα να σκέφτομαι πώς να διατυπώσω την άποψή μου για το μέλλον της Ευρώπης. Το μέλλον της Ευρώπης είναι κάτι που το έχουμε στα χέρια μας, χειροπιαστό. Και θα πρέπει υπεύθυνα να κινηθούμε και για το παρόν και για το μέλλον. Σήμερα το πρωί έγινε συζήτηση στην αλλαγή του κλίματος και συζητήσαμε κάτι που θα είναι χρήσιμο για το μέλλον. Αλλά είναι υποχρέωσή μας για τις μελλοντικές γενιές να κάνουμε κάτι. Και να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι καλύτερο μπορούμε ούτως ώστε να βρούμε εφαρμόσιμε αποτελεσματικές λύσεις που οι λαοί της Ευρώπης θα κατανοήσουν και που θα θέλουν να εφαρμόσουμε. Τι σημαίνει αυτό, να αντικατοπτιστούν οι ανάγκες των λαών, Οι λαοί λένε ότι δεν τους αρέσει η ανασφάλεια και η αστάθεια, την οποία συναισθάνονται. Πρέπει να τους πούμε την αλήθεια. Ξέρω ότι η αλήθεια είναι μια λέξη που δεν την εφαρμόζουν στην ουσία πάρα πολλοί πολιτικοί. Η αλήθεια μπορεί να εκλειφθεί σαν σχετική έννοια. Όμως, πρέπει να υπάρχουν κάποιες σταθερές, σταθερές λέξεις και έννοιες που θα είναι πυλώνες, να υπάρχουν κάποιες αρχές επί των οποίων στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας πυλώνας είναι η αλήθεια. Πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο γιατί κάνουμε κάτι όταν το κάνουμε. Ε, τρομοκρατία, μετανάστευση, αλλαγή του κλίματος, ε, αλλαγές τεχνολογικές τάχιστες αντιμετωπίζουμε, ρατσισμό, εξτρεμισμό. Υπάρχει κατάλογος απειλών και κινδύνων. Ολόκληρος κατάλογος. Και βλέπουμε ότι κάποια από αυτά είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά ευρωπαϊκά. Βέβαια και πολλά προβλήματα προέρχονται έξωθεν. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα δύο είδη κινδύνων. Ε, έχουμε ισχυρότερε αρμοδιότητε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που, όπω σα είπα, τα παράγουμε εμεί. Και να βελτιώνουμε την αντιμετώπιση, αν μα εμπιστευτεί ο κόσμο να το κάνουμε αυτό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και του έξωθεν κινδύνου, την αβεβαιότητα, την αστάθεια στον κόσμο. Να βρούμε μια συνταγή για να χειριστούμε του εξωτερικού κινδύνου. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Πιστεύω ότι αυτή είναι η συνταγή. Να συμφωνούμε επί εφικτών λύσεων. Όλα τα κράτη-μέλη, όλοι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του λαού, όλοι οι δημοκράτες που είναι και θα είναι, ελπίζουμε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άνθρωποι με επιρροή, σε συνεργασία με τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να είναι μια ολιστική προσέγγιση, να συμπεριλαμβάνονται όλοι για να βρούμε λύσεις για το μέλλον. Δύσκολο το έργο. Δύσκολο να χειριστούμε τους εσωτερικούς κινδύνους και τις εξωτερικές απειλές. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά πιστεύω ότι οι πολιτικοί δεν έχουν τον έλεγχο, τον πλήρη της κατάστασης. Ίσως το φαντάζομαι έχουμε τον ψηφιακό χώρο από πάνω το κεφάλι μας, την ψηφική σφαίρα, όπου εκεί δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα που λειτουργεί και λειτουργεί εναντίον μας αυτή η ψηφιακή νέα πραγματικότητα. Πολλέ νέες δυνάμει θεωρούν ότι ο ψηφιακό τομέα, η ψηφιακή σφαίρα είναι ανεξέλεγκτος χώρος, χωρίς νόμου, ζούγκλα που επηρεάζει και δημιουργεί και ζούγκλα στην καθημερινή ζωή. Έχω ένα έγγραφο που μου τα γράψανε καλά και ωραία, αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Μιλάω απ' έξω. Θέλω να μιλήσω για τι επικείμενε εκλογέ, όχι μόνο τι ευρωεκλογέ. Όλε τι εκλογέ που θα θέλαμε να διεξαχθούν στην Ευρώπη, να είναι δίκαιε όλε και έτσι να υπάρχει πλουραλισμός πολιτικός και αυτόνομη λήψη αποφάσεων από πλευράς ε, των ε, ψηφοφόρων. Οι επόμενες εκλογές λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεκινώντας με τις ευρωεκλογέ, δεν θα είναι συνηθισμένε εκλογές. Έχουμε νέους κινδύνους, νέες άπειλες, νέες περιστάσεις. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι. Ένα κίνδυνο είναι η κατάχρηση των ιδιωτικών δεδομένων των ανθρώπων. Κάποιοι θα μας πούν ότι έχουμε μανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία της ιδιωτικότητα. Αυτό βέβαια ο καθένας έχει δικαίωμα στην άποψή του. Θα θυμηθείτε για το GDPR, τη συζήτηση που κάναμε. Τι κάναμε στην περίπτωση Facebook και Cambridge Analytica που ξέσπασε το Μάρτι φέτος. Ήταν σαν να βλέπω ταινία επιστημονικής φαντασίας εφιαλτική. Κάποια εταιρεία λοιπόν, κάποιος οικονομικός παίκτη διείσδησε και απέκτησε τα ιδιωτικά στοιχεία κάθε ανθρώπου. 87 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν θύματα αυτού. Κάποιος μπήκε στον ιδιωτικό τομέα και καταχράστηκε ιδιωτικούς παράγοντες ε, που καθορίζουν ένα ελεύθερο άτομο. Τα στοιχεία αυτά. Τα καταχράστηκαν τα στοιχεία για προεκλογική εκστρατεία, για πολιτικούς σκοπούς. Το συνηθίσαμε αυτό σε, στον εμπορικό κόσμο, στι διαφημίσει κλπ. Όλοι είμαστε στόχοι αυτή τη προσέγγιση. Στον ψηφιακό κόσμο είμαστε υπό το, κάτω από το μικροσκόπιο. Μα ομαδοποιούν, μπαίνουμε σε ομάδες, κατηγορίες και έτσι μπορούν οι διάφορες εμπορικές εταιρείε και εμπορικοί φορείς να μας στοχεύσουν. Είναι εμπορική χειραγώγηση. Αν δεν θέλω όμως να συμμορφωθώ με αυτό. Αυτό είναι διαφορετικό με τη διαφορά να προσπαθούν να με επηρεάσουν, να εκλέξω κάποιου συγκεκριμένου ανθρώπου σε συγκεκριμένα κόμματα κλπ. Και, και με πιέζουν. Άλλο να αγοράζω πράγματα και άλλο να ψηφίζω. Εγώ ψηφίζω για τον πρόεδρο κάποιας χώρας με μεγάλη επιρροή. Δεν ξέρω, ίσως να είμαι αφηρημένη, να τα λέω κάπως αφηρημένα. Αυτή είναι η απειλή που διαβλέπω. Και αυτό το είδαμε στην περίπτωση της Cambridge Analytica. Μπορεί να στοχεύσει επακριβώς κάποιους ανθρώπους να πάρει τα δεδομένα και βάσει των δεδομένων με κλεμμένα δεδομένα μπορεί να επηρεάσει στην εκστρατεία, την προεκλογική. Δεν πάμε μιλάμε τότε για νόμιμες, ανοιχτές και δίκες ε, εκλογές και ότι έχουμε εγγυημένο πολιτικό πλουραλισμό. Αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος η προστασία των ιδιωτικών στοιχείων των δεδομένων. Δεύτερον, ψευδείς ειδήσει, ε, παραπληροφόρηση, χειραγώγηση της κοινή γνώμης. Τρίτος, κινδύνος, κυβερνοασφάλεια και κυβερνοαπειλές και κυβερνοεπιθέσεις. Είπα ότι οι εκλογές ε, δεν είναι, είναι κάτι συνηθισμένο για αυτούς τους οργανώνουν εκλογές ε, με αυτά που προείπα όμως αλλάζει η κατάσταση. Πρέπει να διοργανωθούν κατάλληλα οι φορείς οργανωτικοί για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για είναι κανονικέ εκλογέ. σω να αλλάξει και η νομοθεσία, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει νομοθετική εξουσία, εξαρτάται τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Και πρέπει να είναι έτοιμοι αυτοί που οργανώνουν τι εκλογέ ε, να εξασφαλίσουν ότι οι εκλογέ θα, θα διεξαχθούν με τρόπο που εγγυάται τον ε, πολιτικό πλουραλισμό και την ε, αυτόνομη ψήφο. Στο εκλογικό πακέτο το οποίο σας περιγράφω Θέλουμε πραγματικά να υπάρχει ε, πολιτικός πλουραλισμός, δεξιά, αριστερά, κέντρο, ανεξάρτητη, πρέπει να υπάρχει πλουραλισμός. Όλοι να έχουν δίκαιη πρόσβαση στους ψηφοφόρους. Ε, συστήνουμε να εισαχθούν κανόνες για προεκλογική εκστρατεία στο διαδίκτυο, για θεμητούς κανόνες, διότι όλο και πιο πολύ πολιτική εκστρατεία κινείται στο διαδίκτυο, προς το διαδίκτυο. Δεν θέλουμε καμία λογοκρισία, Δεν θέλουμε διόρθωση ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρηση. Επεξεργαζόμαστε ορισμό παραπληροφόρηση που είναι η σκόπιμη διάδοση πληροφοριών με πρόθεση να, αλλάξει, να αλλάχθει κάτι κρίσιμο. Κάτι πάνω κάτω, δεν έχουμε μπροστά μου τον ορισμό. Το εκλογικό αυτό πακέτο είναι κάτι που περιμένουν τα κράτη-μέλη να το λάβουν σοβαρά υπόψη του. Είναι βάση για συνεργασία. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να καλύψουν και τις τρεις απειλές που περιέγραψα και θέλουμε να δημιουργήσουμε και ένα δίκτυο. Δίκτυο που θα κινείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να καλούμε τα κράτη-μέλη να διορίσουν εκπροσώπους για αυτό το δίκτυο, για να συνεργαστούν μαζί μας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με αυτό το θέμα. Σας είπα ότι οι αρμοδιότητές μας όσον αφορά τον εκλογικό τομέα είναι πολύ περιορισμένοι είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ανήκει στην κυριαρχία των κρατών μελών. Έχουμε ισχυρότερη αρμοδιότητα για την προστασία των δεδομένων, αληθεύει αυτό. Αλλά φανταστείτε ότι η εκλογική διαδικασία υποστεί μίας. λόγω ε, καταχρηστικών και χειραγωγικών τεχνικών ε, σε δύο-τρία κράτη-μέλη μέσω διαδικτύου. Τότε όλη η Ευρώπη θα έχει πρόβλημα αν συμβεί αυτό σε δύο-τρει χώρε και μόνο. Ακόμα και μόνο σε δύο-τρει ασυμβεί θα έχει πρόβλημα η Ευρώπη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα. Είναι το βασικό θέμα τη σημερινή συζήτηση που αφορά το μέλλον της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Χαίρομαι που μπορούμε να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων. Αυτά είναι πολύ επίκαιρα θέματα, πολύ ενδιαφέροντα. Κυρίως αναφερόμενοι στι νέε τάσει, νέου κινδύνου, νέε προκλήσει που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Να κλείσω εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μαζί θα είμαστε θέση να χειριστούμε του κινδύνου και να βγάλουμε την Ευρώπη από αυτή την κρίσιμη ιστορική στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε και εμείς. Σίγουρα θα μας ε, βοηθήσουν οι προτάσεις σας και σκέψεις σας ενώπιση των εκλογών. Τώρα περνάμε στους φίλους μας από το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Ράνολ Λοπατκά πρώτα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ κυρία Χούμπνερ πρώτα απ' όλα για την πρόσκλησή σας σε αυτήν την συνάντηση της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής για να συζητήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Όσον αφορά το σχέδιο έκθεσή σας για το μέλλον της Ευρώπης, μα ικανοποιεί μεγάλο μέρος της έκθεσης, αλλά όχι ολόκληρη. Η σχέση ανάμεσα στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι αναφέρεται στην έκθεση. Και θα σας εξηγήσω αργότερα τι εννοώ. Υπάρχουν προκλήσεις που δεν μπορούν να λυθούν από τις χώρες ε, μέλη. Πρέπει βέβαια να αντιμετωπιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στηρίζω επίσης το ευρωπαϊκό σχέδιο και ότι τα ωφέλη του πρέπει να ε, κοινωνηθούν καλύτερα στον κόσμο. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί καλύτερα για αυτά τα ωφέλη και αυτό σε όλες τις χώρες μέλη. Το Αυστριακό Κοινοβούλιο εδώ και 10 χρόνια πρέπει να ξέρετε ότι έχει εργαστήρια για τη δημοκρατία που απευθύνονται σε νέους, σε οικογένειες υπέρ της δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενημερώνουμε για όλες τις πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10.000 νέοι συμμετέχουν κάθε χρόνο και συμμετέχουν και βουλευτές από όλα τα κόμματα που εδρεύουν στο Κοινοβούλιο. 100.000 νέοι έχουν τη δυνατότητα να είναι σε επαφή με τους βουλευτές και να ενημερώνονται. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ένα κοινό σημείο μεταξύ τους. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από ένα μόνο θεσμό από μόνο του. Χρειάζεται συνεργασία ανάμεσα το ευρωπαϊκό, το εθνικό, το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο. Αυτή είναι μια αναγκαία προϋπόθεση για να έχουμε θετικές εξελίξεις όσον αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο και προκειμένου να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Τα εθνικά κοινοβούλια εδώ έχουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Επιπλέον ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον τα εθνικά κοινοβούλια, επιπλέον από το ευρωπαϊκό βέβαια, αναλάβουν τους ευρωπαϊκούς στόχους, συζητήσουν τις επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτών, ε, πολιτικών και τον αντίκτυπο που έχουν αυτές πάνω στους πολίτες. Η Αυστρία δεν έχει δικαίωμα μόνο να ε, συμμετέχει σε συναντήσεις σαν κι αυτή, αλλά γενικότερα στις συζητήσεις που γίνονται στις διάφορες χώρες και πρέπει να συμμετέχουν και οι ευρωβουλευτές εκεί. Να υπάρχει δηλαδή ένας μόνιμος διάλογος με εθνικούς βουλευτές, με ευρωβουλευτές και ο διάλογος αυτός να γίνεται και με τους πολίτες. Πρέπει να αναφερθώ τώρα στην Task Force και την επικουρικότητα. Αναφέρονται συχνά αυτά στην έκθεσή σας όσον αφορά την Task Force. Παρόλο που αποτελείται από εθνικούς βουλευτές, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Επιτροπή, έχει επιπτώσεις σε όλα τα θεσμικά όργανα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δύσκολου καιρού για την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Η ενίσχυση τη Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή από τη μια και από την άλλη μεριά η ενίσχυση των αρχών τη αναλογικότητα και τη επικουρικότητα. Αυτά τα δύο ήταν πολύ χρήσιμα. Δεν αποκλεί βέβαια το ένα το άλλο. Κάθε θεσμικό όργανο πρέπει να εξετάσει την έκθεση της Task Force και να αποφασίσει τι συνέχεια θα δώσει. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει αντίκτυπο σε όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να την κατανοούμε καλύτερα και να σεβόμαστε την επικουρικότητα και την αναλογικότητα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να έχουμε έναν πιο σημαντικό ρόλο τα εθνικά και τα περιφερειακά κοινοβούλια. Κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου ακόμα ε, δεν έχει γίνει. Δεν έχουμε τον Ευρωπαϊκό Δήμο. Αυτό δεν υπάρχει ακόμα. Δεν έχουμε ευρωπαϊκά διαβατήρια, για παράδειγμα, έχουμε εθνικά διαβατήρια. Τα εθνικά κοινοβούλια αποτελούν ε, πραγματική πηγή δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθεί η γνώση αυτή που έχουν συλλέξει τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να μπορούν μέσω μιας πράσινης κάρτας να μπορούν να συνεισφέρουν και όχι μόνο με την κίτρινη κάρτα που τους επιτρέπουμε να συμμετέχουν τώρα. Και δεν είναι η Άγγελα Μέρκεν που πρέπει να τα εξηγεί, όχι, πρέπει να το κάνουν αυτό τα εθνικά κοινοβούλια. Πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν ότι έτσι όπως κάνει business η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω την αίσθηση, μπορεί και να κάνω λάθος, αλλά έχω την αίσθηση ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μερικές φορές αγνοούν την πραγματικότητα. Και όμως η επικουρικότητα είναι στοιχείο κλειδί υπάρχει στη συνθήκη του Μάστριχτ και στη συνθήκη της Λισαβόνας. Τα εθνικά κοινοβούλια έτσι απέκτησαν πιο ουσιαστικό ρόλο. Όμως δεν τηρήθηκαν πλήρως υποσχέσεις. Αυτή την αρχή της επικουρικότητας πρέπει να την εφαρμόζουμε σωστά. Η καταξιουσιοδότηση πράξης είναι σε αντίθεση ουσιαστικά με την επικουρικότητα. Τώρα έχουμε πάρα πολλέ, πάνω από 140. Αλλά αυτό είναι λάθο. Γιατί δεν μπορεί να μιλάμε από τη μια με τη, για την επικουρικότητα και από την άλλη μεριά να δρούμε με κατεξουσιοδότηση πράξη. Χρειάζεται λοιπόν μια αντικειμενική ανάλυση για να ξέρουμε τι είναι αυτό που θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή συμμετείχα και εγώ σε αυτήν την task force, θα σας πω ποιες είναι οι παρατηρήσεις μου. Πρέπει η Επιτροπή σας, όχι απλώς να σημειώνει την παράγραφο 9 του σχεδίου έκθεσης της Tax Force, εγώ είμαι πεπισμένος ότι η έκθεση της Task Force συνεισφέρει στις μελλοντικέ συζητήσεις όσον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να βλέπει τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια σαν έναν ισχυρό εταίρο ότι είναι ένας τρόπος για να έρθει η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της. Και αυτό νομίζω ότι φαίνεται και με αυτή την έκθεση. Με αυτήν. Αλλά εσείς θα αποφασίσετε τι θα κάνετε με αυτήν. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στον Κρίστιαν Πούχμαν. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα την επιτυχία στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα μέλλον όπου όχι μόνο να στηρίζουν οι πολίτες της δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να έχουν και εμπιστοσύνη σε αυτές. Πιστεύω ότι είναι σημαντικές δύο πτυχές. Το να λαμβάνονται οι αποφάσεις στο κατάλληλο επίπεδο και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει πιο κοντά στους πολίτες, όπως ήδη αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες. Ποιο βρίσκεται πιο κοντά στου πολίτε από τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Πρέπει να ενισχυθεί ο δημοκρατικό έλεγχο ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που κυρίω μπορεί να γίνει μέσω ε, των κοινοβουλίων ε, και τα εθνικά κοινοβούλια, πέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποτελούν σημαντικό παράγοντα στο θεσμικό πλαίσιο. Ο Ζαν Κλοντ Ιούγκερ στην ε, περσινή του ομιλία παρουσίασε φιλόδοξο σχέδιο για το μέλλον της Ευρώπης ε, και ε, έξι σενάρια για μια πιο ενωμένη και πιο δημοκρατική Ευρώπη. Ο πρόεδρος Ιούνκερ επίσης είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ένα δημοκρατικό άλμα προς τα μπρος. Το να γίνει πιο δημοκρατική η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι πρέπει να αυξηθεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Αυστριακού Συμβουλίου θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες πτυχές που έχουν να κάνουν με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιο μεγάλη εμπλοκή, η πιο μεγάλη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις εθνικές υποθέσεις είναι απαραίτητη και ως μέλος εδώ και πολλά χρόνια της ε, Επιτροπής των Περιφερειών ε, και πρόεδρος της Επιτροπής ΕΚΟΝ, θα ήθελα να πω ότι είναι αποτελεί κλειδί για την ε, ολοκλήρωση, για την της Ευρώπης ο ρόλος των τοπικών αρχών. Στην Αυστρία, όπως και σε πολλά άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά θέματα λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη από την πολιτική σε όλα τα επίπεδα και από άλλους ενδιαφερομένους. Ε, ε, από, άλλους ενδιαφερομένους. Και είμαστε πολύ ε, ενεργός παράγοντας στην εκπόνηση γνωμοδοτήσεων και στην παροχή συμβουλών σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο πάντα παρακολουθούσε την ε, πάντα βρισκόταν στην κορυφή όσον αφορά ε, τις ε, ιεραρχήσεις ε, που είχαν να κάνουν με την επικουρικότητα. Επίσης, ε, είχαμε οργανώσει διάσκεψη στη Βιέννη για την επικουρικότητα. Η επικουρικότητα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Αυστρίας, όπως ανέφερε και η κυρία Υπουργό. Στηρίζουμε τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και προσπαθούμε να γίνονται όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά οι εργασίε. Η Αυστρία λοιπόν ε, βρίσκεται σε θέση να συμβάλλει σημαντικά στη σημαντική συζήτηση. Παρακολουθούμε τις ε, συζητήσεις και τον διάλογο που γίνεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημαντική προϋπόθεση όμως γι' αυτό είναι η κοινή κατανόηση, η κοινή ερμηνεία της αρχής της επικουρικότητας. Ε, και ο κύριος Ολοπάτκα το ανέφερε αυτό τα τελευταία χρόνια. Μας ε, δείχνουν ότι πρέπει να δούμε και τις δύο πλευρές του νομίσματος. Υπάρχουν τομείς πολιτικής όπου ε, πρέπει να επιδιώξουμε τη ε, μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων ε, και να κάνουμε πίσω ένα βήμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ υπάρχουν άλλοι τομεί όπου πρέπει να επιληφθεί η Ευρώπη όπω είναι η προστασία των συνόρων, η ψηφιοποίηση κλπ. Επικουρικότητα πρέπει να σημαίνει λιγότερη Ευρώπη εκεί όπου δεν έχει νόημα, δεν έχει να παίξει σημαντικό ρόλο η Ευρώπη, αλλά περισσότερη ευρωπαϊκή συμμετοχή στα θέματα που μπορούν να λυθούν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επικορικότητα και η αναλογικότητα είναι σημαντικές αρχές. Τα κρατήδια της ε, Αυστρίας ε, έχουν δικά της κοινοβούλια, έχουμε και το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο και ε, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τα κοινοβούλια της χώρας σχετικά με τις νομοθετικές πράξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τους δίνει τη δυνατότητα να σχολιάσουν. Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο λοιπόν λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Κοινοβουλίων των Κρατηδίων ε, για να διαμορφώσει τη θέση του. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η, πιο, ε, ε, η αυξημένη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Για να αυξήσουμε το ρόλο στο μέλλον των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιε προκλήσει και κάποιοι στόχοι. Η συνεργασία και ο συντονισμό μεταξύ των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων καθώ και μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αυξηθεί ο ρόλο των περιφερειακών κοινοβουλίων. Θα πρέπει επίση να εξετάσουμε την αύξηση των αρμοδιοτήτων των Εθνικών Κοινοβουλίων με μια πιο προορατική προσέγγιση. και μάλιστα με εμπλοκή του περιφερειακού επίπεδου και των τοπικών αρχών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Κρίστιαν. Τον Λούκα Ζυγή να καλέσω. Έχουμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής εδώ και του δίνουμε το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε πρόεδρε. Thank you so much, uh, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, κυρία πρόεδρε, για την πρόσκληση. Αγαπητή επίτροπε, αγαπητή κυρία Υπουργέ, Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Αθηνικού Κοινοβουλίου, με τα χαρά συμμετέχω σε αυτήν την επίκαιρη συζήτηση, κυρίω μετά την ε, δήλωση του κ. Γιούνκερ για την κατάσταση στην Ένωση, όπου εκεί μίλησε για το σεβασμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και την ανάγκη για ευρωπαϊκό πατριωτισμό. Πολλοί από εσά, αυτή την αίθουσα παρόντε, εκπροσωπείτε τα εθνικά σα ε, κοινοβουλία και οι περισσότεροι από εσά θα έχετε κρίσιμο ρόλο διαμορφώνοντα το αφήγημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση του επόμενου μήνε. Για πολλά χρόνια, και αυτό ισχύει και σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε από διπομπέως τράγο για όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την αδυναμία να αντιμετωπιστούν τεράστιε προκλήσει που εμφανίζονται τάχιστα. Η κυρία Επίτροπο αναφέρθηκε για κοινωνικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, τεχνολογικά, δημογραφικά, γεωπολιτικά προβλήματα και σχετικέ ε, τροποποίησει και αλλαγέ. Τώρα πρέπει να βασιστούμε στα γεγονότα και όχι σε εικασίε που δυστυχώ είναι κάτι που αναφέρεται εκτενέστερα στου πολιτικού λόγου σε πολλέ εθνικέ συζητήσει. Η Ευρώπη μα έδωσε 70 χρόνια ειρήνης και θα μπορούσε να συνεχίσει να μας δίνει περισσότερη ευημερία και ειρήνη αν συνεργαστούμε επικοδομητικά και υπεύθυνα και ο καθένας να παίξει το συγκεκριμένο του ρόλο. Σας διαβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υπήρξε ενεργός προωθητής της συζητήσεως για το μέλλον της Ευρώπης, όπως και στην έκθεση Ρατόντο αναφέρεται. Κάτι που άκρος ε, διακαώς καλωσορίζαμε το Δεκέμβριο του 2015, θετήσαμε μια έκθεση της οποίας ήμουν εγώ κατόπιν ετοίμαστε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητήσατε εσεί, κυρία Πρόεδρε, κυρία Χούμπνερ, για να συμβάλλουμε στην όλη διαδικασία τη εκθέσεως Μπροκ Μπρεσό ε, του Κοινοβουλίου για θεσμική εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι μπορούμε να επανεβεβαιώσουμε το βασικό προβληματισμό που αναφέρατε στην έκθεση για το μέλλον τη Ευρώπη. Δηλαδή, υπάρχει ανάγκη η Ευρώπη, η αυριανή, να βρει μια νέα ισορροπία μεταξύ πιο ανοιχτή Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει δυνατότητε που μπορεί να δημιουργεί ευκαιρίε και απ' την άλλη μια Ευρωπαϊκή Ένωση που φροντίζει, περιθάλπη ε, και φροντίζει με ενισχυμένη διάσταση συμμετοχή. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα τη νομοδοτήσεώ μα τότε. Τρει βασικέ γραμμέ. Καλύτερη εκμετάλλευση τη υφιστάμενη συνθήκη τη Λισαβόνα στου τομεί πολιτική, να ενισχύσουμε την Ευρωζώνη και να ολοκληρώσουμε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών μέσω καλύτερη χρήσεω τη αρχή τη επικουρικότητα που δεν είναι μόνο κάθετη αλλά και οριζόντια. Και πλήρη εφαρμογή του άρθρου 11 περί συμμετοχικής ε, δημοκρατίας. Το 2017 λάβαμε από τον πρόεδρο Γιούνκερ... να παρουσιάσουμε σκέψεις και προτεραιότητες κοινωνίας των πολιτών σαν αφορά τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης. Και η ΕΟΚΕ ήταν ο πρώτος θεσμός που ξεκίνησε διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συζητήσεις για το θέμα στα 27 κράτη-μέλη. Υιοθετήσαμε μια πολύ ιδιαίτερη μεθοδολογία διαβουλεύσεις, διότι οι πολίτες συμμετέχουν στη διαβούλευση για πολλές στρατηγικές. Και το Ευρωβαρόμετρο πολύ συχνά δίνει χρησιμότατα στοιχεία. Επιλέξαμε να έρθουμε σε επαφή με, το, με τους λαούς μέσω των εκπροσώπων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα κράτη-μέλη ε, και προσπαθούσαμε να βρούμε ισορροπία μεταξύ συνωστοσών των εθνικών κοινωνιών των πολιτών στα διάφορα κράτη-μέλη. Και μετά αυτή τη συζήτηση, σε αυτή τη συζήτηση που συμμετείχαν χιλιάδες εκπροσώποι εκπρόσωποι συγγνώμη, και ηγέτε οργανώσεων θετήσαμε ένα ψήφισμα για τη Λευκή Βίβλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μέλλον τη Ευρώπη τον Ιούλιο του 2017. Κάτι που παραθέτεται και αναφέρεται στην Επιτροπή σα. Και το Μάιο του 2018 η ΕΟΚΕ ήταν ο χώρο όπου ε, δώσαμε απαντήσει. Θέλαμε να εκφράσουν την άποψή του. με πάνελ των πολιτών, το διοργάνωσε αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν προώθηση και παρένεση του Προέδρου Μακρόν και του Συμβουλίου και υποδεχτήκαμε πολίτες από όλη την Ευρώπη για να συζητήσουμε. 12 ερωτήσεις θέσαμε για μια διαβούλευση στο διαδίκτυο. Δυστυχώς δεν ήρθαν τα αποτελέσματα μέχρι τώρα, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε άκνες προσπάθειες. Τελικά η ανταπόκριση δεν υπήρχε τόσο ευρύ, όσο ελπίζαμε. Αυτό το πάνελ των πολιτών κάλυψε πέντε ε, τομεί στη διαβούλευση. Βασικό ερώτημα ποιο ήταν. Δεν θα σε εκπλήσει αυτό, είμαι σίγουρος Δημιουργία θέση απασχόληση. Διαφύλαξη του κοινωνικού ιστού, μετανάστευση, περιβάλλον και ασφάλεια καλύψαμε. Οι πολίτες μας απογοητεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατανοούν οι περισσότεροι όμως ότι η εθνική διάσταση δεν είναι το δεδειγμένο επίπεδο για λύση για πολλά από τα σημερινά προβλήματα. Γι' αυτό παράλληλα η δυσαρέσκεια αυξάνεται αλλά και η προσδοκία παράλληλα αυξάνεται εναντί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θέλουν δράση για κάποια θέματα οι πολίτε, Αλλά ένα ξεκάθαρο, ανεξάρτητα από το μέλλον της Ευρώπης, τους επόμενους μήνες, θα δούμε πολλά από τι εκλογέ. θα πρέπει το μέλλον να καθοδηγείται με πρώτη στη μέρημνα για τους πολίτες. Δηλαδή, στο θεσμικό μόρφωμα που θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2018, ο μηχανισμό συλλογή πληροφοριών από πλευρά Συμβουλίου, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβουλίου δεν είναι κάτι που πρέπει να βελτιωθεί αποκλειστικά, αλλά να ενισχυθεί και να υπάρχει καλύτερη διάθρωση τη συλλογή των απόψεων των πολιτών. Το πώ εξετάζουμε σε θεσμικό επίπεδο πρέπει να απαντήσουμε πρώτα απ' όλα όχι στο πώ, αλλά στην εξή ερώτηση. Πώ εξασφαλίζουμε το ότι οι πολίτε θα αισθάνονται ότι είναι στο επίκεντρο και θα είναι στο επίκεντρο του εγχειρήματο. Είμαστε το μέσο μια αλλαγή ε, πάρα πολύ εύκολη η πρόσβαση στι πληροφορίε. Όλα τα σχέδια ε, ψηφισμάτων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι στο διαδίκτυο. Μπορεί κανεί να συμβάλλει, να εκφράσει άποψη, να έχει λόγο. Ταυτόχρονα ο κόσμο πιστεύει ότι υπάρχει αυξανόμενη απόσταση μεταξύ θεσμικών οργάνων και λαού. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα συλλογικό προβληματισμό για το θέμα αυτό. Και θα πρέπει να δούμε πώ να έχουμε πρόσβαση προ τη νεολαία και πώ η Ευρώπη μπορεί ξανά να γίνει ελκυστική για του νέου. Στην αρχή της, παρουσία, της προεδρίας μου, εδώ και μερικούς μήνες, επί τη ευκαιρία της 60 η επαιτίου της Επιτροπής μας, τον περασμένο Μάιο, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για πραγματική αναγέννηση. Ανααναγέννηση την αποκαλώ εγώ. Για να αποθήσουμε την αναγέννηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί Ευρωπαίοι έχασαν το κοινό ιστό, το κοινό αφήγημα. Δεν αισθανόμαστε ότι ανήκουμε σε αυτό το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω όμω ότι είμαστε σε μια στιγμή κρίση που η κρίση μπορεί να οδηγήσει σε μια πραγματική αναγέννηση. Αυτή η ανα αναγέννηση μπορεί να καθοδηγηθεί μόνο από νέε ιδέε. Η παιδεία, ο πολιτισμό, η δημιουργικότητα, η αλληλεγγύη και ο διαπολιτισμικό διάλογο πρέπει να είναι στο επίκεντρο τη προσπαθία. Όπω αναφέρθηκε, υπενθυμίσαμε τη Λισαβόνα. Η φανταστική ιδέα θα πρέπει να γίνει πάθο, συνέστημα, είναι πρόκληση. Πώ να θεσπίσουμε νομοθεσία, να καλύπτουμε ευαίσθητη χρήση τη συνθήκη τη Αβώνα και των σχετικών διατάξεων και αυτέ οι αξίε να μπουν στο επίκεντρο τη προσπάθεια, να τι προστατεύσουμε τι αξίε. Σήμερα μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε με τα εθνικά κοινοβούλια που παίζουν ζωτικό ρόλο, διασυνδέοντα την Ευρώπη με την πολιτική συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να είσαστε οικοδομικοί λύθοι του μέλλοντο τη Ευρώπη. Και υποστηρίζουμε πλήρω ισχυρότερη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια τα επόμενα χρόνια. Είναι σίγουρο ότι το χρονοδιάγραμμα των επομένων μηνών θα είναι κρισίμου σημασία. Έχουμε τέλος Μαρτίου το Brexit, έχουμε μετά 9 Μαΐου Σύνοδο Κορυφή και μετά τέλος Μαΐου ευρωεκλογέ. Ανεξάρτητα από τι ιδέες που έχουν τα θεσμικά μας όργανα, μεγάλες ιδέες, μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω αυξήσεως της δημοκρατική συμμετοχή των ψηφοφόρων στι εκλογέ του Μαΐου. Για να συμβεί αυτό, Όλοι έχουμε ένα καθήκον. Να υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Όχι μόνο για τα προβλήματα τα σημερινά, αλλά για αυτά που πέτυχε τα τελευταία 70 χρόνια. Διότι ακόμα και σήμερα η Ευρώπη είναι ο, καλύτερος τόπος να ζει κανείς και να εργάζεται. Μπενίνι. Όπως είπε και ο Μπενίνι πριν από λίγες μέρες. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι το καλύτερο εγχείρημα για να δωρήσει τα παιδιά σου. Το καλύτερο δώρο για τα παιδιά σου. Κάθε πρόγραμμα και εγχείρημα μπορεί να βελτιωθεί. Πρέπει να αποφύγουμε υπεύθυνα να χάσουμε και τα αυγά και τα πασχάλια. Και τα αυγά και το καλάθι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι προσβλέπουν αυτοί απ' έξω προς εμάς. Εξακολουθούν να μας βλέπουν σαν ένα ενίο καινοτόμο μοντέλο περιφερειακή ενοποίηση που έδωσε ειρήνη και πρόοδο σε μια ήπειρο που σπαράχθηκε επί δύο αιώνε από πολέμου. Σε μερικέ εβδομάδε έχουμε την εκατοστή επέτειο του τέλου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπήρξε μια πάυση μεταξύ των δύο πολέμων, ο Μεσοπόλεμο. Λοιπόν, εν κατακλείδη, πάω στο θεσμικό πλαίσιο τώρα. Τέσσερα πράγματα έχω να πω. Πρώτο, πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου είναι κρίσιμο ο διάλογο. Χρειάζεται διαθρωμένη διασύνδεση με τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είναι ένα τρόπο να εξισορροπήσουμε και κάποιε υπερβολέ και υπερβάσει που λαμβάνουν χώρα στη δυναμική του Συμβουλίου. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι είναι κρίσιμο σημασία να υπερασπιστούμε, να προστατεύσουμε και να διαφυλάξουμε το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τρίτον, πιστεύουμε ότι όσον αφορά το Συμβούλιο πρέπει να σπρώξουμε για περισσότερη χρήση της ειδική πλειοψηφία και να διαβεβαιώσουμε ότι αυτά που αποφασίζονται πρέπει να υλοποιούνται και να γίνει κάτι κανονικό. Μετανάστευση, Φερρυπίν, ασφάλεια, όταν συζητάμε αυτά τα θέματα. Όταν συζητάμε για τη Λιβύη, ό,τι και αν συζητάμε. Από τη στιγμή που παίρνουμε μια απόφαση, αφού τα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να ανταποκριθούν. Και να μην αλλάζουν μετά άποψη και να επαναχωρούν Τέλος, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε πιο διαθρωμένη εμπλοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΟΤΑ και της κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων αυτών μέσω του ρόλου των δύο συμβουλευτικών επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με άλλα λόγια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εστέ βεβαία ότι θα εξακολουθούμε να είμαστε ισχυρό σύμμαχό σα για να διαφυλάξουμε την Ευρώπη των επομένων 60 και να την προθίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου τη Επιτροπής των Περιφερειών τώρα, κυρία Ντούντεν. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά, κυρία Πρόεδρε, είναι πιο εύκολο για μένα, βλέπετε. Κυρία Χύπνερ, αγαπητοί συνάδελφοι από την Επιτροπή ΑΦΚΟ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω στο όνομα του Καλχάιντς Λάμπερτς ε, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την σημερινή πρόσκληση. Δυστυχώ ο, ο κύριος Λάμπρεξ δεν μπορεί να είναι παρόν ε, σήμερα. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια σχετικά με αυτά που υπόθηκαν πριν, ε, σχετικά με την Task Force, ε, την ειδική ομάδα εργασία. Νομίζω ότι είναι σημαντικά για τη συζήτηση αυτή. Η Επιτροπή των Περιφερειών στην Task Force ζήτησε η διαδικασία νομοθεσία στο Συμβούλιο να γίνει πιο διαφανής κάτι που και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι μεγάλης σημασίας. Μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια η Επιτροπή των Περιφερειών ανέλαβε το καθήκον να ε, ευαισθητοποιήσει σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο σχετικά με το θέμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε στην Task Force. Ελπίζουμε όμω εμεί, η Επιτροπή των Περιφερειών, από κοινού να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα συμπεράσματα τη ε, έκθεση αυτή. Θα ήθελα όμω να πω και λίγα λόγια σχετικά με το μέλλον τη Ευρώπη. Η συζήτηση για το μέλλον τη Ευρώπη ε, πράγματι αποτελεί κεντρική πρόκληση σήμερα περισσότερο από ποτέ, όχι μόνο με, υπό το φως ε, των ευρωεκλογών του χρόνου σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και επιτόπου στις πόλεις και στις περιφέρειες, οι ιδέες της ε, Ευρώπης είναι ζωντανοί. Ε, αλλά στους πολίτες διαδίδεται όλο και περισσότερη η αβεβαιότητα, κάτι που εκμεταλλεύονται οι λαϊκιστές όλων των ειδών. Το σχέδιο έκθεσης ε, του συναδέρφου δείχνει ότι πρέπει να ξανασκεφτούμε την Ευρώπη και θα μπορούσε να πει κανείς ότι ναι, χρειαζόμαστε νέες ιδέες. Δεν χρειάζεται όμως να επανεφεύρουμε την Ευρώπη. Τα όσα ήδη έχουμε οικοδομήσει είναι καλά και πολλές από τις αντιφάσεις που συχνά κατακρίνονται ως αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι μάλλον η δύναμή της. Διότι μόνο με συμβιβασμού μπορούμε να συνεργαστούμε και αυτό απαιτεί χρόνο, υπομονή, ενέργεια. Δημιουργεί όμως και τη βάση για αμοιβαία εμπιστοσύνη, κάτι που νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ σήμερα όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η κοινωνία των πολιτών, οι εθνικές κυβερνήσεις, ε, τα πολιτικά κόμματα, ε, οι επιστήμονες, ε, άνθρωποι του πολιτισμού υποβάλλουν προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί η Ευρώπη να γίνει πιο διαφανής και πιο δημοκρατική και μεταξύ άλλων με τους ε, ε, ε, διαλόγους πολιτών που πραγματοποιούνται σε διάφορα μέρη. Η Επιτροπή των Περιφερειών επανειλημμένα έχει ζητήσει οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμμετέχουν πιο ενεργά στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης διότι έχουν, τη καλύτερη, έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν καλύτερα τους πολίτες και να τους κινητοποιήσουν υπέρ της Ευρώπης μπορούν να εξηγήσουν καλύτερα ποιε λύσεις είναι δυνατόν να βρεθούν εντό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ποιες ε, δεν ενδείκνυνται για λήψη αποφάσεων σε αυτό το επίπεδο. Είναι καλύτερα σε θέση να πραγματοποιήσουν ε, επικοδομητικές ιδέες και νομίζω ότι αυτό είναι προς όφελος όλων. Η Ευρώπη των πολιτών είναι η Ευρώπη του μέλλοντος και ε, αυτό αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής των Περιφερειών ε, για το παρόν διάστημα. Θέλουμε να ανανεώσουμε τη σχέση της Ευρώπης με τους πολίτες της ε, και να έχουμε πραγματική ανταλλαγή απόψεων ε, και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σύμφωνο απολύτες, απολύτως μένα από τα συμπεράσματα της έκθεσης που ζητάει περισσότερη διαφάνεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, στη βάση της οποίας να μπορεί να αναπτυχθεί η δημοκρατία. Συμμερίζομαι επίσης και τη θέση ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία απαιτεί ευρωπαϊκή ταυτότητα περισσότερη συμμετοχική δημοκρατία και λιγότερα εθνικά πλαίσια. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι φυσικά ότι αυτά τα στοιχεία πρέπει να αναπτυχθούν ε, ταυτόχρονα. Μόνο αποφασιστική δράση ε, με πολιτική ευθύνη μπορεί να τα φέρει αυτά. Οι δημοκρατικές δομές ε, κατέχουν κεντρικό ρόλο και θα πρέπει να φροντίσουμε όλες οι ευρωπαϊκές αποφάσεις ε, να έχουν τοπική διάσταση και οι τοπικές αποφάσεις να έχουν πάντα ευρωπαϊκή διάσταση θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επικεντρωθεί σε αποφάσεις που να μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών. Συγκεκριμένα έργα για περιφερειακή ανάπτυξη, μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας, ε, ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασφάλιση των ανθρώπων σε έναν ολοένα και πιο χαοτικό κόσμο. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω κάποιες ενέργειες της Επιτροπής των Περιφερειών. Χθες ο πρόεδρος Λάμπερτ μαζί με τον ε, πρόεδρο Ταχάνη, με παρουσία του πρόεδρου Ταχάνη, ε, έκανε την ομιλία του για την κατάσταση της Ευρώπης και οι δύο πρόεδροι δεσμεύτηκαν για συνεργασία διότι αν θέλουμε να πείσουμε τους πολίτες της Ευρώπης ε, και να προστατεύσουμε την το, τολμηρό εγχείρημα της Ευρώπης από την καταστροφή ε, θα είναι απαραίτητη η συνεργασία. Χρειάζεται λοιπόν να οικοδομήσουμε πάλι την εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, κάτι, μια έκκληση την οποία έκανε και ο πρόεδρος Τούσκ. Θα πρέπει να αναλυθούν ε, ευθύνε και από τις τοπικέ αρχές και αυτό ισχύει και για την ένταξη των ε, προσφύγων για παράδειγμα αλλά και για την καταπολέμηση της αλλαγή του κλίματος. Ε, πάνω από 170 μέλη τη Επιτροπής των Περιφερειών είχαν διαλόγους με τους πολίτες και πάρα πολλοί πολίτε συμμετείχαν σε αυτού είτε απευθεία, είτε επιγραμμικά. Επίσης, ε, χιλιάδε πολίτες απάντησαν σε επιγραμμικό ερωτηματολόγιο και έχει αναπτυχθεί εφαρμογή κινητού τηλεφώνου ε, για την υποβολή ιδεών σχετικά με την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν μπορούν να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις ε, για να συνεχιστεί ο διάλογος ε, και μάλιστα όχι μόνο πριν ε, τις ευρωεκλογές και χωρίς ανταγωνισμό σε σχέση με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αλλά ως συμπλήρωμα αυτής. Θα πρέπει όμως επίσης να διασφαλιστεί αυτοί που συμμετέχουν στον διάλογο αυτόν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το τι έχει γίνει με τις ιδέες που έχουν υποβάλει. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε τις επαφές με την κοινωνία των πολιτών ε, που εκπροσωπούνται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Εμείς λοιπόν τα μικρά θεσμικά όργανα μπορούμε να αναπτύξουμε ιδέες και να τις δοκιμάσουμε, τις οποίες θα μπορούμε να ε, υποβάλουμε στα ε, άλλα θεσμικά όργανα και που θα μπορέσουν να φανούν χρήσιμα. Προσβλέπουμε λοιπόν στην ε, ανταλλαγή απόψεων μέσα στους επόμενους μήνες, αλλά φυσικά και μετά τις ευρωεκλογές. Διάλογος, εμπιστοσύνη, εγκύτητα. Αυτά είναι σημαντικά και ο διάλογος οδηγεί στην εμπιστοσύνη συχνά ε, οι πολίτες έχουν εμπιστοσύνη στις τοπικές αρχές τους. Η Ευρώπη θα πρέπει παντού να αποδείξει ότι βρίσκεται κοντά στον πολίτη. Θα πρέπει λοιπόν να αναλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσει σε τοπικό επίπεδο προγράμματα ανταλλαγών, ε, συναντήσεις με άλλους πολίτες ε, είναι από τα πιο ισχυρά επιχειρήματα ε, υπέρ της Ευρώπης. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι δημοκρατική και να δεσμεύεται για τις κοινέ μας αξίες. Θα πρέπει με συνεργασία και με εμπιστοσύνη να σημειώσουμε πρόοδο. Έτσι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ντούντεν. πριν περάσουμε στους ευρωβουλευτές και τους εθνικούς βουλευτές, έχουμε τον κύριο Αλμούνια που είναι εμπειρογνώμονας μας ε, και αυτός. Οπότε θα ήθελα να το ζητήσω να πάρει και αυτό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε στη συνάντηση αυτή τόσο ενδιαφέρουσα για όλους τους Ευρωπαίους, όχι μόνο για μας που βρισκόμαστε εδώ. Άκουσα τις ιδέες των προλαλισσάντων και επιτρέψτε μου εμένα τώρα να σας πω πώς εγώ βλέπω τη συζήτηση και τον προβληματισμό για το μέλλον της Ευρώπης. Το να προβλέψει κανείς το μέλλον φυσικά είναι αδύνατον πόσο μάλλον στους καιρούς που ζούμε. Όμως, είμαστε υποχρεωμένοι, δεδομένων των προκλήσεων ακριβώς που αντιμετωπίζουμε, είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να διευκρινίσουμε ποιες είναι οι ιδέες μας, τουλάχιστον για το τι θέλουμε εμείς για το μέλλον μας, για το μέλλον των παιδιών μας και των επόμενων γενεών. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι και πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Το ευρωπαϊκό σχέδιο αντιμετωπίζει προβλήματα. Εγώ δεν θυμάμαι παλιότερα τέτοιες συζητήσεις για την ίδια την ουσία του ευρωπαϊκού σχεδίου σαν και αυτές που έχουμε σήμερα ε, σε πολλές από τις χώρες μας. Και σίγουρα είναι κάτι που θα συζητηθεί πολύ πριν από τις ευρωεκλογέ. Σε εθνικό επίπεδο, στις χώρες μας ή τουλάχιστον σε πολλές από αυτές, έχουμε προβλήματα με τις δημοκρατίες μας. Όχι μόνο γιατί είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σαν εθνικές δημοκρατίες έχουμε προβλήματα τα οποία πριν από μερικά χρόνια νομίζαμε ότι είχαμε λύσει. Ακόμα και σε πιο νέες δημοκρατίες όπως τη δικιά μου τη χώρα, για παράδειγμα. Έχουμε όμως ταραχές και σε τοπικό επίπεδο και σε παγκόσμιο. Έτσι λοιπόν οι πολίτες μας βρίσκονται με πολλές αβεβαιότητες, με πολλές ανησυχίες. Και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είμαστε αντιμέτωποι με αυξανόμενη πόλωση των κοινωνιών και των πολιτικών συζητήσεων. Οι δύο πόλοι λοιπόν διχάζουν τους πολίτες. Υπάρχουν αυτοί που φοβούνται το μέλλον και υπάρχουν από την άλλη μεριά εκείνοι που φοβούνται το κίνδυνο να πάνε πίσω. Υπάρχουν αυτοί λοιπόν που φοβούνται να πάνε πίσω και γι' αυτό θέλουν να οικοδομήσουν ένα περισσότερο ασφαλές μέλλον. Οι πολίτες ψάχνουν για προστασία ο καλύτερος τρόπος όμως να προστατεύσουμε τους πολίτες ως πολιτικοί, Ευρωπαίοι, υπεύθυνοι, ηγέτες τέλος πάντων, ο καλύτερος τρόπος έλεγα είναι να προσφέρουμε μια καλή προστασία για ένα καλύτερο μέλλον, όχι για να πάμε πίσω. Συζητάμε λοιπόν για το πώς θα το κατορθώσουμε αυτό. Υπάρχει δημόσιος χώρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο Κάποιος είπε μάλιστα στην αρχή σήμερα το απόγευμα ότι δεν υπάρχει Ευρωπαϊκός Δήμος. Πράγματι, ακόμα δεν έχουμε πετύχει τον Ευρωπαϊκό Δήμο, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και των επόμενων που ακολούθησαν μέχρι σήμερα, συμμετέχουμε σε όλο και περισσότερο ευρωπαϊκές συζητήσεις που έχουν κοινού παράγοντες σε όλες μας τις χώρες. Ποιοι συμμετέχουν στις συζητήσεις? Τα κοινοβούλια, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τα εθνικά κοινοβούλια συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση και γι' αυτό είναι πολύ χρήσιμε τέτοιε συναντήσει. Συμμετέχουν επίση τα πολιτικά κόμματα, περισσότερο βέβαια σε εθνικό επίπεδο παρά σε ευρωπαϊκό. Θεσμικά τα κοινοβούλια έχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαν συνομιλητή, ενώ τα πολιτικά κόμματα δεν είναι τόσο ισχυρά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να γίνονται και σε τέτοιο επίπεδο θεσμικές συζητήσεις. Και βέβαια όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο γίνονται τέτοιες συζητήσεις, στην κοινωνία των πολιτών και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από παλιά. Είναι πιο δύσκολο σήμερα να υπάρξει ένας ηγέτης από ό,τι πριν από κάποιες δεκαετίες. Γι' αυτό και είναι πιο δύσκολο να συνεχίσουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Λείπουν οι ισχυροί ηγέτες, ηγέτες που να μπορούν να εγκαθιδρύσουν διάλογο και όχι βέβαια ηγέτες που να θέλουν να επιβάλλουν. Αυτό είναι το σημείο κίνησης για τον προβληματισμό μας. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, ποια είναι τα δύο κύρια κεφάλαια στον προβληματισμό αυτό για το μέλλον της Ευρώπης. Από τη μια μεριά έχουμε τις θεσμικές πτυχές. Και εδώ θα μπορούσα σε λίγα λεπτά να σας πω ποιες είναι οι δικές μου οι ιδέες για τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που πιστεύω ότι χρειάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάβασα την έκθεση που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο σας, από αυτού, και σίγουρα θα μελετήσω προσωπικά και την επόμενη έκθεση του αγαπητού φίλου Χαουράκη. Εγώ δεν πιστεύω ότι θεσμικές αλλαγές πρέπει να γίνουν επιγόντως τώρα με αλλαγή της συνθήκης. Κάποια μέρα εντάξει θα αλλάξουν πάλι οι συνθήκες, αλλά προς το παρόν οι θεσμικές αλλαγές που έχω εγώ στο μυαλό μου δεν χρειάζονται. Μην ξεχνάμε ότι το 2005 απέτυχε η συνταγματική συνθήκη και θυμάμαι επίσης και την αποτυχία της Νίκιας και τότε που προσπαθήσαμε δηλαδή να προετοιμάσουμε το έδαφος. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα θεσμικά στα περιθώρια των τωρινών συνθήκων, χωρίς να χρειάζονται δηλαδή αλλαγές στις συνθήκες. Είμαι υπέρ του να χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη πασαρέλ, που δεν χρησιμοποιήθηκε μετά τη Λισαβόνα. Είμαι υπέρ επίσης της ενισχυμένης συνεργασίας. Έχουμε τέτοια παραδείγματα ενισχυμένης συνεργασίας μέχρι σήμερα, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε η μέθοδος αυτή να χρησιμοποιείται περισσότερο, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρούμε χωρίς να αναβάλουμε αλλαγές, επειδή δεν μπορούμε να πετύχουμε ομοφωνία στο Συμβούλιο. Θα συμφωνήσω, και το είπατε κι εσείς, ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι βέβαια θεσμικό όργανο στη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά πιστεύω ότι έχει υπερβολικά πολλές εξουσίες. Η υπερβολική επιρροή, η θεσμική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βρήκε την καλή ισορροπία από τη στιγμή που θεώρησε θεσμικό όργανο το Συμβούλιο. Εγώ αναγνωρίζω την ανάγκη να υπάρχουν στρατηγικές συμφωνίες και στραγικοί προσανατολισμοί από τους ηγέτες μας, τους επαφαλείς κρατών κυβερνήσεων, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε πώς θα τηρεί την νομοθεσία, πώς θα εφαρμόζεται, ποιος ε, θα παίρνει τις αποφάσεις και τι αποφάσεις ακριβώς. Όλα αυτά στα χέρια του Συμβουλίου είναι υπερβολικά. Έπειτα έχουμε το θέμα τη ειδική πλειοψηφία που δεν υπάρχει σήμερα στο Συμβούλιο, χρειάζεται ομοφωνία. Και αυτό έχει τι συνέπειε. Το αναβάλλονται έτσι πολύ σημαντικέ αποφάσει. Πρέπει το θεσμικό μας πλαίσιο να λειτουργεί πιο ομαλά, άρα με περισσότερες αποφάσεις, με ειδική πλειοψηφία και για τα φορολογικά και για θέματα αγορών. Πρέπει να χρησιμοποιείται η κοινωτική μέθοδος περισσότερο από ό,τι διακυβερνητική και πρέπει επίσης να ενισχύσουμε το διάλογο ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Το είπαν και άλλοι πριν από μένα και συμφωνώ απόλυτα με τέτοιες ιδέες. Τώρα, τι μπορούμε να πετύχουμε με τις θεσμικές αυτές αλλαγές. Θα σας δώσω πέντε σημεία πολιτικών που κατά τη γνώμη μου χρειάζονται αποφάσεις για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρώπη από εδώ και πέρα και να μην αναβάλουμε αυτή τη βελτίωση για αργότερα. Λοιπόν, πρώτον, να ολοκληρωθεί η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Δεν θα μπω εδώ σε λεπτομέρειες. Είναι γνωστοί οι οδικοί χάρτες, έχουν συζητηθεί ξανά και ξανά και εδώ και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Χρειαζόμαστε διορθώσεις σε θέματα διακυβέρνησης της Οικονομικής Ένωσης. Οι Υπουργοί της Ευρωζώνης πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτό πρέπει να δούμε τις καλές σχέσεις επίσης, αυτών που είναι εντός και των εκτός, δηλαδή όταν οι Βρετανοί δεν θα βρίσκονται πια εδώ. Η εκτός μπορεί να είναι μια μειοψηφία, αλλά τα μέλη της ε, Ευρωζώνης δεν θα πρέπει να αγνοούν τις σκέψεις, τις ανησυχίες, και τις επιθυμίες των υπολείπων που είναι εκτός της Ευρωζώνης. Πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτοί που δεν είναι έτοιμοι να μπουν στο ευρώ δεν πρέπει να πιεστούν και να το κάνουν στα γρήγορα. το Κοινοβούλιο της Ευρωζώνης δεν θα πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτό εδώ το Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω ότι πρέπει να βρει τον τρόπο να εξετάσει τα θέματα της Ευρωζώνης χωρίς να χωριστεί στα δύο. Και πρέπει επίσης να δώσουμε περισσότερη προσοχή και έχει το δικαίωμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει αρμοδιότητες για τις συζητήσεις που γίνονται όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για την Τραπεζική Ένωση, δεν πρόκειται μόνο για την ε, ικανότητα την ε, δημοσιονομική, πρόκειται και για τη σύγκληση, πρόκειται για την ανταγωνιστικότητα, πρόκειται για την καινοτομία, πρόκειται για την απασχόληση, πρόκειται για την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Όλα αυτά απαιτούν πολύ σημαντικές συζητήσει και όχι μόνο σε επίπεδο του Συμβουλίου μεταξύ Κομισιών και Συμβουλίου ή σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων και των ε, αρμόδιων επιτρόπων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει με τα εθνικά κοινοβούλια και να παρακολουθούν την τήρηση των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να ζητήσουν αρμοδιότητες για εκείνες τις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια που δεν τηρούν τις συστάσεις που αποτελούν ένα κοινό αγαθό για όλους τους Ευρωπαίους και όχι μόνο για αυτούς που υποφελούνται πιο άμεσα. Πρέπει να συζητήσουμε βέβαια και για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική που δεν υπάρχει. Και αυτό το θέμα μαζί με την τρομοκρατία είναι τα θέματα που περισσότερο απασχολούν τους πολίτες μας. Και εφόσον ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Δεν έχουμε όμως προχωρήσει καθόλου όσον αφορά μια κοινή μεταναστευτική πολιτική. Και όμως οι πολίτες μας περιμένουν να είμαστε εμεί στην πρώτη γραμμή. Να μην, να μην αγνοούμε βέβαια την αρχή της επικουρικότητας, αλλά να ηγηθούμε των αποφάσεων για ένα τόσο καυτό ζήτημα για τους πολίτες μας, που μπορεί να αποτελέσει και κίνδυνο για την ίδια τη δημοκρατία μας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται πολιτικό σθένος, πολιτική ηγεσία, πολιτική βούληση, αλλά αυτό σημαίνει ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια ότι πρέπει να συμμετέχουν στις συζητήσεις που γίνονται για τις μελλοντικέ προκλήσεις Χρειάζεται ηγετικός ρόλος, χωρίς βέβαια να επιβάλλονται οι ιδέες. Χρειάζεται δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Σήμερα η δημοκρατία είναι μια πολυεπίπεδη πρόκληση για όλους μας. Το θέμα δεν είναι αν υπάρχει έλλειμμα δεξιά-αριστερά εδώ-εκεί, όχι. Έχει να κάνει με όλα τα επίπεδα των πολιτικών μας δράσεων. Άρα Χρειάζεται να ξαναβρούμε, να ανοικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρώπη, η οποία μειώθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει κάποια πρόοδος τελευταία ορισμένες χώρες, επειδή σταμάτησε η ύφεση και αρχίζει και πάλι μια νέα θετική προοπτική όσον αφορά την ανάπτυξη. Όμως η εμπιστοσύνη είναι κάτι αναγκαίο για την Ευρώπη. Χωρίς την εμπιστοσύνη των πολιτών η Ευρώπη δεν έχει μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Ακή. Έχω λάβει μόνο 10 ονόματα από εκείνους που θέλουν να λάβουν το λόγο. Υπάρχει άλλος? Για να μοιράσουμε το διαθέσιμο χρόνο. Στο επόμενο πεντάλεπτο, αν αποφασίσετε θέλετε να μιλήσετε, πείτε το μας. Πριν σταθώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, Λιθουανία πρώτα. Μιντάουγκας Πουίντικας από το Βίλνιους, από το Κοινοβουλίο. Έχετε το λόγο. Pone pirmininkė, kolegos, iš tiesų Lietuva nuoširdžiai nori, kad ES projektas. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Λιθουανία θέλει το ευρωπαϊκό εγχείρημα να είναι επιτυχές. 64% των πολιτών των, της χώρας μας υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν εργάστηκα σαν εμπειρογνώμονα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2014, κατέγραψα σαφώς τα προβλήματα που θα αντιμετώπιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit ήταν μόνο ένα από τα πολλά προβλήματα και ήταν, θα έλεγα, συναγερμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στου πολλού συναγερμού που σήμαναν. Πρέπει να συζητήσουμε την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Αυτό είναι ένα θέμα που μα διχάζει. Θέλουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα να είναι μακρόπνοο, συνεχέ, επιτυχέ. Αν θέλουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να θυμόμαστε την αλήθεια που ο κ. Στόμχαν, ο Βρετανός ιστορικός, εξέφρασε. Είπε λοιπόν ο Βρετανός ιστορικός ότι διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις εμφανίζονται στον πολιτικό κόσμο όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Βασική απειλή που αντιμετωπίζουμε είναι η διάλυση, η αποσύνθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνεται αντιληπτή σαν ένωση ισοτήμων κρατών μελών που ενώνονται από Όσον αφορά ξεχωριστά ζητήματα, μπορούμε να δούμε ότι η χώρα μας ενδιαφέρεται όσον αφορά την αποφυγή διεθνών υπερεθνικών καταλόγων ψηφοδελτίων για τις ευρωεκλογέ. διότι έτσι δεν εξασφαλίζεται η επαρκής ευθύνη και δεν είναι σωστή επιρροή στι ευρωεκλογέ. Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και θέματα δημοσιονομικά, είναι πολύ σημαντική επικουρικότητα. Επέκταση της ειδική πλειοψηφία. Εκεί βλέπουμε ότι στη δήλωσή του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ, πρότεινε η ειδική πλειοψηφία να εφαρμόζεται στον τομέα Τη φορολογίες και σε άλλου τομεί με κάποιες εξαιρέσει. Αυτές οι πτυχέ πρέπει να συζητηθούν, διότι οδηγούν σε φεντεραλισμό και έτσι τα μικρότερα κράτη-μέλη στερούνται της δυνατότητας να εισακουστούν. Τούτου λεχθέντος πρέπει να πω ότι 64% του πληθυσμού μας είναι υπέρ της Ευρώπης και στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλέ πολλές δείχνουν ότι ο κόσμος δεν αισθάνεται ότι εισακούει τη φωνή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να προβούμε σε μία ανάλυση. Ανάλυση των προτάσεων των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Πολύ συχνά αυτές οι χώρες λένε ότι δυτικοευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να επιβάλλουν το δικό τους θεματολόγιο, τη δική τους ατζέντα. Οι χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και οι πολίτες αυτών των χωρών δεν θέλουν να θεωρούνται ε, πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Θα πρέπει κάθε κάτος μέλος να έχει φωνή που εισακούεται. Για να λαμβάνονται αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές οι αποφάσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικότερες. Να υπάρχει μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία και να συγκεντρωθούμε περισσότερο ε, στα προβλήματα της κοινωνίας. Συνάδελφοι, πραγματικά εύχομαι η, αυστριακή, η ουγγρική, η ιταλική φωνή, η σλοβακική φωνή, οι φωνές όλων των χωρών ακούγονται. Πρέπει να βρούμε βιώσιμες λύσεις στον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι θα γίνουμε ισχυροί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Από το Ευρωκοινοβούλιο, ο Λάινεν έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα για τη σημερινή συζήτηση, διότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε μόνο να το διαμορφώσουμε από κοινού. Δεν μπορεί να το κάνει μόνο του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε μπορεί να το κάνει μόνο του κάποιο εθνικό κοινοβούλιο. Αποτελεί κοινό εγχείρημα. Και νομίζω ότι αυτό το είπαν και όλοι οι ομιλητές. Ζήτησα το λόγο διότι δυστυχώς ε, στις 4 ε, ε, πρέπει να πάω να ψηφίσω την έκθεσή μου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για τη διάσκεψη για το κλίμα στο Κάτοβιτ. Ο πρόεδρος Χαβιελούκα είπε ότι έχουμε ξεχάσει γιατί ε, δημιουργήσαμε και γιατί ε, θέλουμε να συνεχίσουμε να διατηρούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Δυτική Ευρώπη κάποια πράγματα μπορεί να είναι ε, να ήταν σαφή κατά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστασία των εξωτερικών συνόρων. Αλλά Ας κοιτάξουμε και την Κίνα και να δούμε τι οικονομική πρόκληση αντιμετωπίζει για μας. Έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό. Ε, δεν είναι ελεύθερη αγορά η Κίνα ε, ε και συχνά τα προϊόντα της Κίνας ε, λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις ε, και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό κανένα ευρωπαϊκό κράτος, ούτε η Γερμανία δεν μπορεί να το κάνει αυτό μόνη της. Ας κοιτάξουμε την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Ξέρουμε ότι καταβάλλονται προσπάθειες, επενδύονται δισεκατομμύρια και στην Κίνα και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Για να διασφαλίσουμε το μέλλον με σύγχρονες τεχνολογίες χρειαζόμαστε ένα κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα, χρειαζόμαστε κοινέ προσπάθειες, ε, χρειαζόμαστε εμβληματικές πρωτοβουλίες. Έχουμε μείνει πίσω όμως, χάνουμε. Ε, και μόνο από κοινού με κοινά ερευνητικά προγράμματα μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Όσον αφορά τη δημοκρατία, η συνθήκη της Λισαβόνας λέει ακριβώς αυτά που θέλουμε. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και έχουμε συμμετοχική δημοκρατία. Όσον αφορά την κοινοβουλευτική δημοκρατία, σύντομα θα έχουμε ευρωεκλογές. Εδώ και 40 χρόνια έχουμε τέτοιες διακρατικές εκλογές ε, ως ε, μόνο μέρος σε όλο τον κόσμο. Και γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό. Δεν ε, θα είχαμε όμως κοινοβουλευτική δημοκρατία αν δεν είχαμε τους απαραίτητους παράγοντες. Δηλαδή, ισχυρά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Αυτά υπάρχουν στο χαρτί. Στην πραγματικότητα όμως δεν υπάρχουν ακριβώς και νομίζω ότι ε, η διαδικασία του candidate, του κορυφαίου υποψηφίου θα είναι καλή διότι για πρώτη φορά θα έχουμε προσωπικότητες, θα παρουσιάζονται προσωπικότητες πέρα από τα εθνικά σύνορα. Και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, θα έχουμε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και μεγαλύτερη προβολή. Την Ευρώπη λοιπόν μπορούμε να την οικοδομήσουμε μόνο από κοινού και θα ήθελα πολύ ε, συμμετοχή των ε, Εθνικών Κοινοβουλίων. Αναφέρατε την πράσινη κάρτα, αυτό θα είναι το επόμενο βήμα μετά την κίτρινη κάρτα. Και εγώ Ήμουν μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών ως εκπρόσωπος ε, της ε, γερμανικής κυβέρνησης και γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η κυρία Ντούντεν ανέφερε την μόνιμη δημιουργία διαλόγου των πολιτών. Συνέχεια δηλαδή μέσα από το τοπικό επίπεδο να συμμετέχουν οι πολίτες. Και ε, Χαβιέρ, πρόεδρε, μου άρεσε πολύ η ομιλία σου και νομίζω ότι ε, είναι ένας από τους καλύτερους ε, τόπους ε, να μένει κανείς η πατρίδα σου και δεν θα επιτρέψουμε να καταστραφούν αυτά. Και αυτό το λέω και σε όλους τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη. Άλλος ένας συνάδελφος πρέπει να πάει... Η Μαργέτε πρέπει να πάει να ψηφίσει. Μήπως θέλει να πάει στο λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τον Μάιο ήθελα να πω ότι είχαμε έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που επέκρινε τη δουλειά στο Συμβούλιο, τόνισε ότι δεν υπάρχει διαφάνεια και ότι δεν ενεργούν με ευρωπαϊκό τρόπο. Ε, οι πολίτες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά που κάνουν οι δικές τους οι κυβερνήσεις. Η Επιτροπή μας, λοιπόν, μαζί με την Επιτροπή των Αναφορών, της οποίας είμαι μέλος, έχουμε μια εξαιρετική έκθεση και ο Λάινεν είναι ένας από τους εισηγητές και απαντάμε στις επικρίσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Σα καλώ λοιπόν, πηγαίνετε στι κυβερνήσει σα, πείτε του ότι πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορά και όχι να φέρονται σαν να είναι διακυβερνητικό φορέα χωρίς διαφάνεια, χωρίς δημοκρατική συμμετοχή, χωρίς ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θα πρέπει να είναι εξίσου διαφανής με εμά εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα πρέπει να μπορείτε να παρακολουθείτε τι κάνει η δική σας κυβέρνηση και πώς συναλλάσσετε με τι άλλε κυβερνήσει, με τρόπο ώστε να αναλάβουν ευθύνη για τις δικές τους αποφάσεις. Η εξαιρετική έκθεση του Γιώ Λάινεν δείχνει ότι ε, όπως έχουν τα πράγματα τώρα μπορούν απλά να κατηγορήσουν τις Βρυξέλλες για ό,τι πάει στραβά. Δεν θα μπορέσουν ποτέ οι πολίτες να συμμετάσχουν σε όλες τις εργασίες εάν δεν φερόμαστε με δημοκρατικό και διαφανή τρόπο. Η κυρία Οράιλη, η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, απαντάει ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς αλλαγή των συνθήκων. Πρέπει να αλλάξει κανείς συμπεριφορά και νοοτροπία. Αλλά μπορούν έτσι να περάσουν σε άλλο τρόπο εργασίας, ώστε να συμμετέχουν και τα εθνικά κοινοβούλια στη διαδικασία αυτή και να έχουμε πολύ πιο αξιόπιστες μεθόδους εργασίες από τις πράσινες, κόκκινες κάρτες κλπ. Σας καλώ λοιπόν να ακολουθήσετε αυτή τη γραμμή. Και σας παραπέμπω στην, εθνική, στην ειδική έκθεση της διαμεσολαβήτριας. Θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα. Και έχουμε και εμεί σε σχέδιο έκθεση τη Επιτροπή Αναφορών και τη Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Έχει ημερομηνία 1η Ιουλίου και έχει αριθμό 2096. Θα ήθελα λοιπόν να συστήσω σε όλους να διαβάσετε αυτά τα δύο έγγραφα. Έτσι θα έχετε στα χέρια σας ε, καλά εργαλεία για να αναγκάσετε τις κυβερνήσεις σας να ενεργήσουν με τρόπο διαφανή και αξιόπιστο. Αυτό θα βοηθήσει όλους μας και στην επαφή με τους πολίτες μας ώστε να καταλάβουν πώς μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο αναλαμβάνοντας τις δημοκρατικές τους ευθύνε ε, χωρί να λένε απλά ότι α, δεν μπορούμε διότι είναι όλα πολύ επικίνδυνα, είναι πολύ μακριά από εμά κλπ. Ευχαριστούμε πολύ. Ραμόν, Ραμόν Χωράγκη τώρα για να παρουσιάσει την εκθεσή του. Και ευχαριστούμε που περιμένατε τόσο υπομονετικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ειλικρινά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπορούμε να σχολιάσουμε σε βάθος και να μιλάμε μεταξύ μας ειλικρινά, να ανταλλάσσουμε απόψεις για το πώς βλέπουμε την Ευρώπη και το μέλλον της. Γιατί δεν είναι όλα ίδια και πρέπει να το ξέρουμε αυτό και να το αναγνωρίζουμε. Ευχαριστώ την Αυστριακή Προεδρία, το Κοινοβούλιο ε, της Αυστρίας, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και φυσικά και το φίλο μου και σύντροφό μου Χωακίμ Αλμούνια ο οποίος κατά τη γνώμη μου έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση. Κάτι που θέλω να πω σε όλους τους βουλευτές και ευρωβουλευτές, να τους πω ότι τους ευχαριστώ πολύ για τη συμβολή τους. Λοιπόν, γιατί μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί. Γιατί βρίσκεται υπό αμφισβήτηση το μέλλον της Ευρώπης. Αυτό είναι το πρώτο που δυστυχώς πρέπει να δεχτούμε. Είμαστε σε μια κρίση που ο ίδιος ο κύριος Γιούνκερ ανέφερε ότι είναι υπαρξιακή. Είμαστε στην άκρη του γκρεμού με τα οικονομικά προβλήματα, με την κρίση του ευρώ, το Brexit, τη μεταναστευτική κρίση, την εσωτερική τρομοκρατία κλπ. κλπ. Δηλαδή η Ευρώπη περνάει δύσκολα χρόνια. Και υπάρχει γενικός προβληματισμός. Πώς να οικοδομήσουμε το μέλλον της Ευρώπης μέσα από αυτή την κρίση. Σε αυτό όμως προστέθηκε και ότι υπάρχει μια γενικευμένη άποψη ότι η Ευρώπη που γνωρίζουμε προχωράει δύσκολα, αργά, ότι σαν υπερεθνικό όργανο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ταχύτητα με την οποία προχωρούν τα συμβάντα με τον ίδιο ρυθμό που προχωράει η πραγματικότητα. Υπάρχουν θεσμικά εμπόδια δηλαδή που εμποδίζουν την Ευρώπη να ανταποκριθεί με την ευελιξία που χρειάζεται στην εξωτερική πολιτική, για παράδειγμα την οικονομική σύγκληση, με το ότι έχουμε την Ευρωζώνη και τους υπόλοιπους. Όλα αυτά βαραίνουν και δυσκολεύουν μια συζήτηση που είναι αναγκαία. Επίσης δημιουργήθηκε στο εσωτερικό μια ένταση μεταξύ των εθνών που ποτέ δεν είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα υπάρχει μια διαφορά βορράς-νότος στη μακροοικονομική πολιτική. Επίσης ένα χάσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης για το μεταναστευτικό που ποτέ δεν είχαμε προηγουμένως. Και γι' αυτό και γίνεται αναγκαία ακόμα περισσότερη συζήτηση και ο προβληματισμός για το μέλλον της Ευρώπης. Πρέπει να δούμε πώς επίσης θα αριθμιστεί το μέλλον όταν θα έχει αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί σίγουρα κατήχε μια σημαντική θέση. Τώρα είμαστε αναγκασμένοι να επαναδιαμορφώσουμε το χώρο αυτό. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησε να προκαλέσει αυτή τη συζήτηση γιατί υπάρχει πεποίθηση ότι ελοχεύουν όλο και περισσότεροι κίνδυνοι και έχουμε όλο και περισσότερες προκλήσεις μπροστά μας που μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν όλοι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, όλοι όσοι ήρθαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχουν αναγνωρίσει όσοι ήρθαν να μας παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης. Ο καθένας μας είναι πολύ λίγος, πολύ μικρός, δεν μπορεί να μένουμε διχασμένοι. Και το εξέφρασε και ο πρόεδρος Γιούνκερ, ότι ό,τι υπάρχει στο οριζοντά μας, εμπορικές σχέσεις, σχέσεις με την Κίνα όπως είπε ο Ζολάινεν, άλλες σχέσεις, εμπορικές πολιτικές κτλ. απαιτούν συνεργασία στο φορολογικό για την αντιμετώπιση των απατών της φοροδιαφυγής, ε, επειδή υπάρχουν ε, η φορολογική παράδεισοι. Έπειτα, οι δημοκρατικές μας αξίες και αρχές Υπάρχει τώρα μια νέα δημοκρατία του διαδικτύου. Εμείς οι Ευρωπαίοι πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, πώς θα συμπεριλάβουμε σε αυτό το νέο σώμα τις αρχές μας, τις αξίες μας, πώς θα πετύχουμε την προστασία των δεδομένων αν δεν έχουμε μια Ευρώπη ισχυρή που να μπορεί να ανταγωνιστεί στα πλαίσια ενός διαδικτύου Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια Ευρώπη περισσότερο ισχυρή που να κάνει μια κοινωνική πολιτική που δεν κάνει. Υπάρχουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι που περιμένουν από την Ευρώπη να ανταποκριθεί, να προσφέρει μια κοινωνική πολιτική. Το θέμα της μετανάστευσης που επήγει. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να το λύσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί είναι ένα πρόβλημα που ήρθε για να μείνει μαζί μας όλο τον 21ο αιώνα. Συνεπώς η πεποίθησή μου είναι εξή. Πώς θα προβληματιστούμε για την Ευρώπη, όχι για να την ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Όπω είπε η πρόσωπο τη Επιτροπή των Περιφερειών, δεν πρόκειται να φτιάξουμε μια διαφορετική υπερεθνική ένωση. Όχι, αλλά πρέπει να υπάρχει ευελιξία, πρέπει να τη βελτιώσουμε την Ευρώπη που έχουμε σήμερα. Και ολοκληρώνω, συνάδελφοι, με κάτι που δεν θέλω να είμαι προκλητικός, απλώς θέλω να τονώσω τον προβληματισμό. Συχνά ακούμε, ακόμα και από κάποιο πρωθυπουργό το ακούσαμε, εδώ, της Ολλανδίας. Να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα, είπε. Ειλικρινά ρωτάω, μα γίνεται. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με λιγότερους οικονομικούς πόρους, για παράδειγμα. Υπάρχει μια ιδέα που κυκλοφορεί τώρα που ετοιμάζουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε λιγότερους πόρους. 14-15 εκατομμύρια. Αλλά θέλουμε να κάνουμε από την άλλη περισσότερα. Να κάνουμε περισσότερα, τι άμυνα λέμε, για να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, ε, τεχνητή νοημοσύνη, είπαμε ψηφιακά, ενέργεια. Έχουμε τόσες προκλήσεις, τόσα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε. Μα θα τα κάνουμε με λιγότερα, είναι δυνατόν. Εγώ νομίζω πως δεν γίνεται. Αν θέλουμε να κάνουμε περισσότερα, δεν μπορούμε να τα κάνουμε και με λιγότερες νομοθετικές εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούν να γίνουν περισσότερα αν ο κεντρικός άξονος της Ευρώπης είναι το έθνος και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι είναι ασύμβατα αυτά μεταξύ τους. Εγώ είμαι από αυτού που πιστεύει ότι υπάρχουν ε, πολλές κοινέ ταυτότητες. Είμαι Βάσκος, είμαι Ισπανός, Ευρωπαίος. Τι άλλο, α, και από την πόλη μου. Το που ανήκει κανείς μπορεί να ανήκει σε πολλά πράγματα συγχρόνως να έχει πολλές ταυτότητες συγχρόνως. Δεν μπορεί να λέμε ότι ο μόνος χώρος δημοκρατίας είναι το έθνος. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται από 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Εγώ δεν πιστεύω, όπως είπε κάποιος, ότι είναι μια φανταστική κοινότητα. Όχι, δεν είναι καθόλου φανταστική. Είναι μια πραγματική κοινότητα εθνών και πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όμως θέλουμε να μιλήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης. Εξού και το πνεύμα της έκθεσης αυτής. Φυσικά και περιλαμβάνει και την ιδέα ότι φυσικά και χρειαζόμαστε τα Εθνικά Κοινοβουλία. Όλα όσα είπατε τα ακούμε και είναι πολύτιμα και χρειάζονται στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Αναλογικότητα, επικουρικότητα βεβαίως. Τα ακούμε και συμφωνούμε. Αλλά αυτό που λέμε εδώ είναι ότι η απουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε διάφορα θέματα που ρυθμίζουν τελικά το Συμβούλιο και Επιτροπή και εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα καν να έχουμε διάλογο νομοθετικό γιατί θέλουν μόνο διαβούλευση μαζί μας και όχι να συναποφασίζουμε, μας αποδυναμώνει. Το είπε και ο κύριος Αλμούνια. Μας απασχολεί λοιπόν Και τελειώνω με αυτό κυρία Πρόεδρε. Όλο και πιο συχνά βλέπουμε ότι δεν τηρείται το ευρωπαϊκό δίκαιο σε πολλές χώρες. Και εδώ δεν μιλάω μόνο για τις ποσοστώσεις μεταναστών. Πολλές φορές το ευρωπαϊκό το κοινοτικό δίκαιο δεν τηρείται από πολλές χώρες και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου που ασχολούνται με τις ανταλλαγές ιατρών μεταξύ των χωρών μας ή προσωπικού με μπλε κάρτα, τέλο πάντων που θα μπορούσε να απασχοληθεί σε διάφορε χώρε, είναι κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψη από πολλέ χώρε. Άρα η ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών δεν γίνεται σεβαστή από πολλέ χώρε. Πολύ σημαντικό αυτό ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο πρέπει να τηρείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλιώς αποδυναμώνεται ολόκληρη η Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ε, ναι, που είσαστε εδώ, συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια, για να μας δώσετε τη γνώμη σας, να προβληματιστείτε μαζί μας. Χρειαζόμαστε ένα ρεύμα ευρωπαϊστικό, που φυσικά και να σέβεται τις αρχές της συνεργασίας, αλλά χρειαζόμαστε ένα ρεύμα που να ζητάει μια περισσότερο ισχυρή Ευρώπη, πιο ισχυρή Ευρώπη, όχι για να κάνει λιγότερα, μια Ευρώπη που να μπορεί να κάνει περισσότερα στα πλαίσια βέβαια του σεβασμού των αρχών μας. Αυτό είναι που χρειαζόμαστε για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ραμόν. Συνάδελφοι, βάσει του καταλόγου που έχω, μέχρι πέντε λεπτά έχει ο καθένας. Αν ζητήσουν κι άλλοι το λόγο, θα πρέπει να αρχίσω να περιορίζω το χρόνο. Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλή των Λόρδων. Ο Λόρδος Λίτλ έχει το λόγο. Ρότζερ, πού είσαι? Ευχαριστώ που με καλέσατε, με φωνάξατε. Αισθάνομαι ντροπή που παρευρίσκομαι με την εγκύτητα του Brexit και λυπάμαι πολύ για την απόφαση που έλαβε η χώρα μας στο δημοψήφισμα. Τι θέλω να σας πω σήμερα. ότι δεν φτάσαμε στο τέλος της ιστορίας. Από το 2016 όλοι αναγνωρίζουν πια ότι η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό που φαντάστηκαν. Δεύτερον, αναγνώρισαν τώρα ότι δεν μπορείς να έχεις και την μπίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Υπάρχουν σοβαρές απώλειες και από πλευράς επιρροής και από πλευράς οικονομικής όταν αποχωρεί κανεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θα συμβεί τι επόμενε εβδομάδες, ιδέα δεν έχω. Υπάρχουν πολλές απόψεις για το τι πρόκειται να συμβεί. Θα ήταν τραγικό αν πιστέψει ο κόσμος ότι η μόνη επιλογή ήταν μεταξύ συμφωνίας που μπορεί να πετύχει στις Βρυξέλλες η κυρία Μέη και καμιά συμφωνία. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών. Υπάρχει πραγματική δυνατότητα μιας πολιτικής κρίσης που μπορεί να ξεσπάσει στη Βρετανία και από αυτή την κρίση ενδεχομένως θα υπάρχει δυνατότητα να σταματήσει το Brexit. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν είναι τη επιτροπή μου ή επιδήποτε άλλου. Νομίζω ότι στη Βρετανία αντιμετωπίζουμε μία από τις πιο έντονες κοινοβουλευτικές περιόδους. Η ατμόσφαιρα είναι ατμόσφαιρα μεγάλης κρίσης που επικρέμεται. Και πραγματικά οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί σε αυτή την ατμόσφαιρα. Τώρα, αν τελικά πραγματοποιηθεί το Brexit, ποια είναι η απόψή μου για τα θέματα που συζητούμε σήμερα το απόγευμα. Πρώτα απ' όλα, ο Βρετανός πρέπει να καταλάβει ότι είναι σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία για να μπορεί να πετύχει και η Βρετανία εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε τόσα πολλά κοινά στοιχεία. Αντιμετωπίζουμε πολλά παρόμοια προβλήματα. Οι αξίες και τα συμφέροντα ε, είναι πάνω κάτω τα ίδια. Και θέλουμε να πετύχει η Ευρώπη. Από την πλευρά μου, και νομίζω ότι αυτό αληθεύει για την ε, γνώμη που στη Βουλή των Λόρδων και στο κόμμα μου, στο εργατικό κόμμα. Πιστεύω λοιπόν ότι αν λάβει χώρα το Brexit, θέλουμε να παραμείνουμε όσο πιο, πιο κοντά γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σε όλες τις πτυχές. Τι σημαίνει αυτό. Να διατηρήσουμε την βαθύτερη δυνατή σχέση με την Ευρώπη να υπάρχει διάλογος σε βήματα όπως το σημερινό. Και η Επιτροπή μας επιθυμεί διακαώς να παραμείνει τμήμα της ευρωπαϊκής συζητήσεως, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί το Μάρτι. Υπάρχει και ένα παράδοξο που σχετίζεται με το δημοψήφισμα περί Brexit. Ποιο είναι αυτό. Για πρώτη φορά, τώρα, στη Βρετανία, υπάρχει φιλοευρωπαϊκό εκλογικό σώμα το ΣΥΠΗΝ. Είναι εκείνοι που ένθερμα θέλουν να είναι στην Ευρώπη. Κυρίως οι νέοι το θέλουν αυτό. Οι νέοι θεωρούν ότι είναι ένα θέμα ταυτότητας. Θέλουν να είναι Ευρωπαίοι. Και πιστεύουν ότι οι παλαιότερες γενναίες ψήφισαν στο δημοψήφισμα για να μειώσουν τις ευκαιρίες που θα έχουν αυτοί στο μέλλον. Θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση με θέμα το τι μπορούν να κάνουν μαζί η Ευρώπη και η Βρετανία για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα των καιρών μας. Όχι μόνο θέματα ασφαλείας, αβεβαιότητα που βρισκόμαστε σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες, με τον Πούτιν, με την τρομοκρατία και όλα τα υπόλοιπα αλλά ποια είναι τα οικονομικά προβλήματα, η αλλαγή του κλίματος. Είναι κάτι που μας επηρεάζει όλους και πολύ. Δημογραφικά θέματα, μετανάστευση, πώς μεταρρυθμίζουμε τον καπιταλισμό ούτω ώστε να γίνει βιώσιμος και να παράγει δίκαια αποτελέσματα για όλους στην κοινωνία μας. Αυτά είναι κοινά ζητήματα. Κοινά ερωτηματικά που αντιμετωπίζουμε ως Ευρωπαίοι και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε και μετά τον Μάρτιο. Και ακόμα εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορεί να παραμείνουμε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που σεβαστήκατε το πεντάλεπτο, αλλά ελπίζουμε ότι αυτή την τελευταία φορά που θα σας δούμε, ότι θα μπορέσουμε, θα πρέπει να σεβαστούμε την απόφαση της χώρας σας, λυπούμεθα για αυτό που συμβαίνει και αυτή η Επιτροπή θα παράσχει τη σύμφωνη γνώμη. Αυτό είναι το παράδοξο. Ότι προσμετρούμε την επιτυχή διαδικασία του Brexit μέσω της επιτεύξεως συμφωνίας βάσει της οποίας θα αποχωρήσετε. Πιθανότατα αυτό θα συμβεί. Και τώρα, καλό, την κυρία Μάλετιτς, μέλος Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, που έχει συνεργαστεί με τον Ραμόν Χουαρέγγι και ετοίμασαν ε, μια σχετική έκθεση. Ε, γνωμοδότηση για την έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλου του συναδέλφου των Εθνικών Κοινοβουλίων και νομίζω ότι είναι πολύ καλό που συζητούμε μαζί για να μπορέσουμε ε, να συμμετέχετε εσείς περισσότερο, διότι εκεί εσείς μπορείτε να εξασφαλίσετε την πραγματοποίηση, την υλοποίηση των πολιτικών στην πράξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ιβάνα, Μπορεί να πλησιάσει το μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Στην Επιτροπή Οικονομικών Μεσμετικών Θεμάτων αποφασίσαμε να παρακολουθούμε στενότερε οικονομικέ πολιτικέ, να παραμείνουμε σε αυτό το θέμα και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι η γνωμοδότηση ήταν μια ευκαιρία να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να υποστηρίξουμε την ολοκλήρωση διαδικασιών που ξεκίνησαν προετών όπως η διαδικασία ολοκληρώσεως της Τραπεζικής Ενώσεως και ανάγκη να εξασφαλίσουμε ανοιχτή προσέγγιση και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση. Να ολοκληρώσουμε και την ε, ενιαία αγορά κεφαλαίων, διότι η εμβάθυνση και ολοκλήρωση αυτού του τομέα είναι κάτι που συμπληρώνει την Τραπεζική Ένωση και θα συμβάλλει στον επιμερισμό του ιδιωτικού κινδύνου, θα αυξηθεί η οικονομική σύγκληση και θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε καλύτερα ε, μελλοντικού κλειδονισμού. Μετά έχουμε τη διαδικασία εμβάθυνση και ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ενώσεως, ούτως ώστε να διαφυλαχθεί η σταθερότητα του ενιού νομίσματος και να αυξηθεί η σύγκληση οικονομικής, δημοσιονομικής, πολιτικής και πολιτικής της αγοράς εργασίας μεταξύ κρατών Τέταρτον, να γίνουν και άλλα βήματα για την ανάπτυξη μηχανισμού σταθερότητας στην Ευρώπη και να έχουμε και το θέμα του Ταμείου ε, ε, Επιλύσεως, μάλλον ρευστοποίησεως τραπεζών και διάσωσης τραπεζών. Όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, ακόμα συζητούν τα κρατη και δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τη δημιουργία αποτελεσματικών και αναλογικών μέτρων για ένα σύστημα ευρωπαϊκό ασφάλειας καταθέσεων και αυτό είναι ένα απομένων ε, πυλώνα τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Και εδώ βλέπουμε και το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μπορείτε να το συζητήσετε αυτό και να προσπαθήσετε να έχετε μια σταθερή θέση όσον αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Τραπεζικής Ένωσης και όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που ανέφερα, ασφάλεια των καταθέσεων. Μετά καλύτερη ε, πρόσβαση στις κεφαλαγορές, θα βοηθά τις νοφυείς εταιρείε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσονται γρήγορα, πολύ σημαντικό και αυτό, και οι παραδοσιακές ΜΜΕ ξέρουμε ότι εξαρτώνται από ε, δανειοδότηση τραπεζών και θα πρέπει να εισαχθούν νέα μέτρα και εγγυήσεις που θα αυξήσουν τη δυνατότητα του τραπεζικού τομέα να δανειοδοτεί περισσότερο προγράμματα μεγαλύτερο κίνδυνο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπούν μεγαλύτερο κίνδυνο. Πρέπει να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε την υλοποίηση συστάσεων αναχώρα, κάτι που συζητήθηκε επανειλημμένα στο Ευρωκοινοβούλιο, μαζί με εσά επίσης, με τα μέλη των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων, πώς να βελτιώσουμε τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και θεωρούμε ότι μεγαλύτερη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων που θα συζητούν εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων εκθέσεις ε, ε, αναχώρα και συστάσεις αναχώρα θα βοηθήσει να τα απορροφήσουν όλα αυτά οι χώρες οπότε θα εφαρμόζουν καλύτερα τις συστάσεις αναχώρα διάφορες χώρες, ενστερνιζόμενε τις συστάσεις Και έτσι θα βελτιωθεί η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι επενδύσει, η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και η εφαρμογή διαφθορτικών μεταρρυθμίσεων είναι οι τρεις πυλώνε για την επίτευξη βιώσιμη ανάπτυξη. Συνεπώ, Υποστηρίζουμε και το μελλοντικό πρόγραμμα InvestEU, επενδύστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επένδυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κάτι ευπρόσδεκτο. Θα αποτελεί συνέχεια το InvestEU του ΕΦΣΥ, του προγράμματος για θετικές επενδύσεις και θα οδηγήσει σε νέες επενδύσεις σε ύψος 38 δις ευρώ. Θα πρέπει να κατευθύνεται σε ιδιωτικά προγράμματα με κίνδυνο, καινοτομία και ταχεία ε, ανάπτυξη των νεοφιών επιχειρήσεων να πω ότι οι ε, μεταρρυθμίσεις χρήζουν υποστήριξη. Υπάρχει σχετικό πρόγραμμα στον τρίτο πυλώνα του τριγώνου. Αυτό το πρόγραμμα ήταν πιλωτικό στι παρούσε δημοσιονομικέ προοπτικέ και ο αριθμό των αιτήσεων για υποστήριξη από κράτη-μέλη ξεπέρασε κατά πολύ τον σχεδιαζόμενο προπολογισμό. Πέρα των επενδύσεων, και τη υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική χρειαζόμαστε και τι διαθωτικέ μεταρρυθμίσει που θα εφαρμόζονται υπεύθυνα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να στηρίξουμε νέε μεταρρυθμίσει και σχετικά προγράμματα υποστήριξη αυτών στο νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει σχετίζεται αυτό με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και εφαρμογή των συστάσεων αναχώρα στα διάφορα κράτη-μέλη πρέπει να στηρίζεται. Τέλο. Πολύ σημαντικό και αυτό. Στη γνωμοδότηση η δημιουργία ενιαίου καθεστώτος για το ΦΠΑ και συστήματος για το ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί πάνω από 25 χρόνια το επεξεργαζόμαστε αυτό. Και ήρθε η ώρα να μειωθεί το κόστος συμμορφώσεων για τις επιχειρήσεις, να μειωθεί ο κίνδυνος διασυνοριακής απάτης στο ΦΠΑ και να πλουστευθούν οι διαδικασίες σχετιζόμενες με το ΦΠΑ, κάτι που θα ενισχύσει την ενιαία αγορά και θα δημιουργήσει καλύτερε συνθήκε για τι επιχειρήσει και διασυνοριακό εμπόριο. Στη γνωμοδότηση τονίζουμε αυτό, ότι θα πρέπει πραγματικά να επιταχύνουμε τη διαδικασία ε, δημιουργίας οριστικού συστήματος ΦΠΑ και χρειάζεται και διαδικασία προσαρμογής του φορολογικού συστήματος, τεχνολογικές εξελίξεις και στην ψηφιοποίηση και θα πρέπει να αλλάξουν τα επιχειρηματικά μοντέλα σύμφωνα με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ιβάνα. Εστονία η κυρία Λόνερ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάθε πρωί που ανοίγουμε τα μάτια μας, βλέπουμε ότι υπάρχει κάποιος Ευρωπαίος πολίτης δυσαρεστημένος. Και αυτό εξαιτία της, ε, όχι τόσο της θεσμικής δομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά περισσότερο εξαιτία της υποκρισίας της ευρωπαϊκής πολιτικής, γιατί η Ευρώπη υπόσχεται προστασία, ευημερία, όμως τελικά λιτότητα προσφέρει και μειώνει τις δημόσιες υπηρεσίες και προκαλεί αβεβαιότητα για το μέλλον. Μετανάστευση, για παράδειγμα. Η δημόσια συζήτηση και οι προτάσεις αγνούν πλήρως το γεγονός ότι η μετανάστευση είναι ένα οικονομικό φαινόμενο. Οι ε, μεγάλες ροές μετανάστευσης χρειάζονται επειδή χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό. Και τελικά καταλήγουμε στο ότι χρειαζόμαστε περισσότερο πληθωρισμό. Άνθρωποι έρχονται από επικίνδυνα μέρη, από επικίνδυνα σημεία του κόσμου, τις περισσότερες φορές για οικονομικούς λόγους. Η Ευρώπη σήμερα εμπλέκεται στο θέμα της μετανάστευσης για κόσμο που έρχεται από κάπου που οι οικονομικές συνθήκες είναι πολύ κακέ. Και εμεί τους κλείνουμε την πόρτα, παρόλο που χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό. Αυτό είναι υποκρισία. Για να σταματήσει αυτή η υποκρισία λοιπόν πρέπει να βρούμε νέες κοινέ αρχές για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την οικονομία που γίνεται περισσότερο παγκόσμια και για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε την ε, αγορά εργασίας που πρέπει να εξυπηρετεί τον κόσμο η μετανάστευση θα σταματήσει στην αγορά εργασίας. Τα σύνορα πρέπει να είναι περισσότερο ασφαλή, αλλά και οι συνθήκες εργασίας πρέπει να είναι περισσότερο ασφαλείς. Τώρα όταν κυρίαρχες χώρες είναι υποχρεωμένες να δεχτούν ποσοστώσεις, δεν μιλάμε για λύσεις. Ακριβώς αυτό είναι το μέρος του προβλήματος, γιατί οι ποσοστώσεις αυτές αποτελούν μία υπόσχεση σε μεγάλες επιχειρήσεις ότι θα έχουν περισσότερο φτηνό εργατικό δυναμικό. Αν λοιπόν θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες όταν ανοίγουν τα μάτια τους το πρωί να σκέφτονται ότι η Ευρώπη είναι καλός χώρος για να ζει, πρέπει να ξαναδούμε όχι τόσο τη δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να υπογραμμίσουμε περισσότερο το θέμα της πλήρους απασχόλησης. Αν κάθε Ευρωπαίος που θέλει να βρει δουλειά, τη βρίσκει, την έχει και όταν έχει δουλειά ξέρει ότι έχει και δικαιώματα εργασιακά, τότε η μετανάστευση θα είναι θέμα ελεύθερης επιλογής και όχι κρίση. Η πλήρης απασχόληση αποτελεί την προϋπόθεση για να συζητήσουμε για οικονομική ανάπτυξη και για ισότιμη ανάπτυξη. Η Ευρώπη έχει μέλλον εφόσον βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών της και οι πολίτες της μπορούν να κάνουν ελεύθερα τις επιλογές τους και να μην είναι μία ένωση στην υπηρεσία των ε, μεγάλων ε, επιχειρησιακών συνασπισμών. Ευχαριστούμε πολύ που τηρήσατε και το χρόνο σας. Ουγγαρία, Σόλταν Σουλντιντέτσι. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να συμμετάσχω στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Υπάρχουν διάφορα σχέδια εκθέσεων που έχουμε εξετάσει τις τελευταίες εβδομάδες. Εμείς πάντα θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη που να αποτελείται από ισχυρά κράτη-μέλη. Αυτή είναι η αφετηρία μας. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε προστασία των συνόρων και σωστή διάκριση των αρμοδιοτήτων. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε μιλήσει και με τα άλλα κράτη Βίσεγκρατ και καταλήξαμε σε μια συνενετική λύση. Όσον αφορά την ασφάλεια ή την ψηφιακή επανάσταση, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Η Ισχυρή Ευρώπη όμως ε, δεν θα έχουμε αν δεν έχουμε ισχυρά εθνικά κοινοβούλια. Ιδιαίτερα θα χαιρόμασταν εάν θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο και περισσότερη επικουρικότητα όσον αφορά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει να σκεφτούμε εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τον ηγετικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επανέλθει στο ρόλο του θεματοφύλακα των συνθήκων. Είναι σημαντική να διατηρήσουμε τα καλά της Ευρώπης και αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε και στο πλαίσιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση Σαρτζεντίνη. Ήταν μεγάλη απογοήτευση, διότι αναφέρθηκαν παλιές παραβάσεις που είχαν ήδη κλείσει και αναφερόταν σε θέματα που αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εάν υπήρχε συνέπεια θα έπρεπε να ε, ε, στυλιτευθούν και άλλα κράτη-μέλη. το Ουγγρικό Κοινοβούλιο αποστασιοποιείται από την επιστολή σε Αργεντίνη για να έχουμε ασφάλεια ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Ε, είναι σημαντικό η Ουγγαρία να λάβει περισσότερους πόρους για προστασία των εξωτερικών σύνορων, που είναι εξωτερικά σύνορα και της Ουγγαρίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεν θα επιτρέψουμε να εισέλθουν λαθρομετανάστες. Προσφέρουμε όμως ανθρωπιστική βοήθεια σε περιοχές όπως είναι η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή. Αλλά ε, δεν θέλουμε να προστατεύουμε τους οικονομικούς μετανάστες. Ευχαριστώ. Τουρκία. Τι Τη Επιτροπή για την Εναρμόνιση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ευχαριστώ πολύ. Ως μέλη της Μεγάλης τουρκική εθνοσυνέλευση χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ σήμερα στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. Πιστεύουμε ότι όλες οι υποψήφιες χώρες πρέπει να καλούνται στην συζήτηση αυτή για να ανταλλάσσουν απόψεις με τους υπόλοιπου για αυτό το θέμα. Ως υποψήφια χώρα Δεν είμαστε σε διαπραγματεύσεις, αλλά έχουμε κληθεί σε έναν προβληματισμό για μετά την συνθήκη της Λισαβόνας. Υπάρχουν πολλές και πολυεπίπεδες προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η Ευρώπη. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις στα προβλήματα αυτά μέσα στο σημερινό κόσμο. Και τα προβλήματα δεν λύνονται από μια χώρα μεμονωμένα. Το βλέπουμε αυτό και με το Συριακό. Οι υποψήφιες χώρες πιστεύουμε ότι μπορούν να βοηθήσουν στην ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και ισχυρή Τουρκία και μια ισχυρή Τουρκία σημαίνει και ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν η Ευρώπη έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Εμείς έχουμε βοηθήσει την Ευρώπη στην προσφυγική κρίση και τις συνέπειές της. Χάρη στη δικιά μας αποφασιστικότητα, μετά τη δήλωση της 18 Μαρτίου έχουν σταματήσει οι ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Βαλκάνια κατά 90%. Συγκεκριμένο παράδειγμα Η, η Τουρκία συγγνώμη, πάντα έχει συνεισφέρει στη σταθερότητα της Ευρώπης και στην ευημερία της. Παρά ό,τι οι αρνητικές σκέψεις υπάρχουν για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς είμαστε υπέρ της ένταξης αυτής. Και χαιρόμαστε που μπορούμε να συνεισφέρουμε στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και τώρα και στο μέλλον. Έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα. Αυτό που έχει σημασία είναι η διεύρυνση. Η Ευρώπη δεν πρέπει να ξεχνάει ότι η διεύρυνση είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση Οπότε η προοπτική της ένταξης χωρίς διακρίσεις μεταξύ των υποψηφίων χωρών είναι κάτι που πρέπει να περισχύσει. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την προοπτική νέων μελών. Όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούγκερ στη συζήτηση για την κατάσταση πραγμάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να παραμείνει μια Ευρώπη των 27. Υπάρχουν ε, υποψήφιες χώρες όπως είναι η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Τουρκία θα μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στις προκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, now we go to Ireland. Ευχαριστώ. Πάμε στην Ιρλανδία. Gerard Crockwell από τη Γερουσία της Ιρλανδίας. Ευχαριστώ κυρία Χούμπνερ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Ευχαριστώ για την αφοσίωσή σα στο όλο εγχείρημα, Πρόεδρε. Έχετε οργανώσει πολλέ τέτοιε συνεδριάσει και το παραδέχομαι. Τώρα, το μέλλον για την Ευρώπη. Ίσως για να το κάνουμε αυτό να ρίξουμε ματιά σε αυτό που είπε ο, ο κ. Χιούμαν. Δεν θα δημιουργηθούν τα πάντα εν μία νυχτή με, βάσει ενό σχεδίου, αλλά μέσω συγκεκριμένων επιτευμάτων που θα δημιουργήσουν μια de facto αλληλεγγύη. Αυτό το μήνυμα είναι σημαντικότατο σήμερα που προχωράμε. Στα 60 χρόνια μετά την έναρξη του εγχειρήματο του ευρωπαϊκού, ξεκινήσαμε από οικονομικό εγχειρήμα προς ένα πολύ ευρύτερο εγχείρημα που καλύπτει πολλές πτυχές της κοινωνικής ζωής. Θα ήλπιζα να μιλούσαμε για 28 χώρες σήμερα, δυστυχώς όμως το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε απόφαση για τον Brexit. Ποιο είμαι εγώ για να μπορέσω να κρίνω η αδίποτε δημοκρατική απόφαση μιας χώρας. Είχαμε παρόμοια εμπειρία και στην Ιρλανδία με τα δημοψηφίσματα. Και ένα τμήμα της ηγεσία το να γείται κανείς τι είναι. Να πας να ξαναρωτήσεις, να ξαναζητήσεις ξανά την άποψη, να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα και να είσαι ειλικρινής έναντι του εκλογικού ε, σώματος. Καμιά φορά θα εκπλαγείς ότι αντιστρέφεται η άποψη του κόσμου. Εγώ στα, από τα συνδικάτα ε, με την κατάλληλη διατύπωση διαπίστωσα ότι τα πάντα μπορεί να τα πετύχει κανείς. Προχωρά η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την επέκταση προ τα Δυτικά Βαλκάνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηρίξει την ειρήνη, ε, θα πρέπει να μάθουν οι χώρες να συμβιώνουν πριν ε, ε, γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην μπαίνουν και να φέρνουν μαζί τους τα προβλήματα. Χαίρομαι που είμαι εδώ, σαν Ιρλανδός εκπρόσωπος μιας χώρας όπου 92%, 92 του λαού σε πρόσφατη έρευνα ήταν αφοσιωμένη όσον αφορά το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Αυτό είναι σημαντικότατο, διότι η λέξη αλληλεγγύη αναφέρθηκε εδώ. Οι Ιρλανδοί δεν είδαν καμία αλληλεγγύη από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα όταν ξέσπασε η χρηματοπιστωτική κρίση και είχαμε 64 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος που επί θα τα ξεπληρώνουμε. Χάρη όμως την ηγεσία των πολιτικών μας και εγώ είμαι ανεξάρτητο γερουσιαστή, δεν μιλώ εκ μέρου κυβερνήσεω ούτε αντιπολιτεύσεω. Χάρη στην ηγεσία μα, καταφέραμε να παραμείνει το πλοίο μα στην επιφάνεια. Να, να, να ανακάμψουμε από την κρίση και να ισχυροποιήσουμε την οικονομία μα, να γίνει ψυχηρότη στην Ευρώπη. Η νέοι είναι το κλειδί. Αν δείτε τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματο του Brexit, οι νέοι δεν ήθελαν να φύγουν από την Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη είναι ο χειρότερο εχθρό τη. Θυμάμαι όταν, με, όταν ήμουν ένα σπουδαστή, μου λέγανε ότι, κάθε φορά ο πελάτη, εγώ σπούδαζα marketing και μου λέγανε ότι όταν κάνει λάθο το μάθουν 10 πελάτε. Ο ένα το πει σε 10. Αν τα πάω καλά, ο ένα ε, θα τα πει σε άλλου τρει. Και δεν το προωθήσαμε το θέμα, δεν κάναμε καλό marketing. Απολαμβάνουν είναι το έρασμο, αλλά δεν σκέφτονται από πού προέρχεται το έρασμο. Οι γεωργοί απολαμβάνουν ε, τα ευεργετήματα τη Γεωργίας Ευρωπαϊκή, αλλά δεν σκέφτονται από πού προέρχονται τα ευεργετήματα. Αλλά όλοι θα σα πούν ότι η Ευρώπη, ότι μας πρόχνει με το ζόρι να υπακούσουμε στον τάδε το δίνα κανόνα, μα υποχρέω να το δεχτούμε. Και πρέπει να κάνουμε κάποια περικοπή όσον αφορά την επιβολή των απόψεων των ε, γραφειοκρατών τη Ευρώπη. Θα πρέπει να εργαστούμε με του ΟΤΑ, με την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι με τα εθνικά κοινοβούλια. Να πλησιάσουν προ τα κάτω να διαθέτουμε, να προωθούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουμε marketing, να, να παρουσιάσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν κάτι υποφελέ για όλου. Μόνο όταν ο λαός καταλάβει τι θα χάσουν, εάν καταρρεύσει το εγχείρημα, τότε θα έχουμε κέρδη. Δεν είναι μόνο τα ε, οικονομικά ωφέλη, αλλά τη παιδεία, τα ωφέλη τη ειρήνη. Όλα αυτά που κερδίζει κανεί αν είναι κομμάτι τη Ευρώπη. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για αλληλεγγύη, α ξαναμπούμε στη σωστή τροχιά, συνεργαστούμε. Ε, είναι μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα μου το Brexit. Αλλά η μεγαλύτερη απειλή, πιστεύω, για όλη την Ένωση είναι το θέμα της μετανάστευσης. Και νομίζω ότι θα χρειαστούμε μια συνεκτική προσέγγιση, στέρεη προσέγγιση και να την προσυπογράφουμε όλοι. Όλοι να αναλάβουν, να υπομισθούν το βάρος τους που τους αναλογεί. Όσον αφορά τα εθνικά κοινοβούλια, με τα χαρά ακούω, άκουσα την ομιλία που ανα... τις ομιλίες που αναφέρουν για καλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. Εγώ θα ήθελα καλύτερη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν θα, ε, επικοινωνίας για τους συναδέλφου του Ηνωμένου Βασίλειου όσον αφορά το Brexit. Ξέρω ότι ελπίζουν για το καλύτερο δυνατό. Εγώ είμαι μέλος ε, μιας λέσχης golf. Ε, Αν δεν πληρώσει τα τέλη δεν μπορεί να παίξει golf στη λέσχη. Δεν θέλω σκληρό Brexit. Δεν θέλω σύνορα στα, στην ίσο τη Ιρλανδία. Πρέπει να βρούμε όμω μια λύση. Και γρήγορα, αρκετά γρήγορα. Διότι ο κόσμο αρχίζει και ανησυχεί. Υπάρχουν πολλοί πρασπιστέ ε, της, ε, του Brexit που μετακίνησαν τι επιχειρήσει του στην ε, Ιρλανδία για να ωφεληθούν από τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκή Πέρασε ο χρόνο μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το χρόνο που με θέσατε. Ευχαριστώ. Ήταν καλό που σα άκουσα. Και ελπίζω να βρεθούν οι κατάλληλε λύσει. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ισπανία. Σοσιαλιστέ. Ερίκε Γκερέρο, έχετε το λόγο. Gracias, eh, Presidenta. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλές λύσεις να προτείνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα. Συμφωνώ πάντως με την Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων στις ε, θέσεις που έχει οθετήσει τα τελευταία χρόνια μέσω εκθέσεων που έχουν ε, εκπονήσει συνάδελφοι Χώσταφ, Μπρόκ, ε, ε, Μπρέσολε και εσείς ίδια ή του Ραμόν Χαγερή που προτείνουν λύσεις για περισσότερη ολοκλήρωση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω να κάνω μερικά σχόλια εγώ μόνο για κάποια προβλήματα που έχουμε, όχι μόνο στην ανατομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στη λειτουργία της. Όχι μόνο δηλαδή στη δομή, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνω 10 χρόνια Ευρωβουλευτής. Προηγουμένως, απέκτησα μεγάλη εμπειρία σε εθνικό επίπεδο. Και η εμπειρία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπίπτει απόλυτα με την δεκαετία της κρίσης που όπως είπε και ο Ραμόν Χιδωρή προηγουμένως δίχασε την Ευρώπη πάρα πολύ. Παλιά λέγαμε ότι η Ευρώπη προχωράει με κάθε κρίση. Όμως αυτή τη φορά πρέπει να πούμε ότι οι κρίσεις βοήθησαν την Ευρώπη να προχωρήσει με αποφάσεις που ελήφθησαν διακυβέρνησης, αλλά τώρα μέσα στην Ευρώπη έχουμε και αντιπαραθέσεις και μπορούμε να πούμε ότι με αυτή την τελευταία κρίση μάλλον πήγαμε πίσω. Μεγάλο μέρος των προβλημάτων μας οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ολοκλήρωση της εθνικής πολιτικής με την ευρωπαϊκή. Και είναι αυτό πολύ σημαντικό να το πούμε τώρα που είμαστε εδώ με εθνικούς βουλευτές και ευρωβουλευτές. Στη συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται ο συνεχής διάλογος ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, λοιπόν, αυτό δεν έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά. Και αυτό φαίνεται σε συναντήσεις σαν και αυτή που έχουμε σήμερα. Φαίνεται δηλαδή η δυσπιστία από τα εθνικά κοινοβούλια προς την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε σε διάλογο μεταξύ μας. Υπάρχει επίσης αυξανόμενη ασυμμετρία ανάμεσα στην ε, πολιτική δράση και στην εκπόνηση των πολιτικών οι πολιτικές έχουν όλο και περισσότερο ευρωπαϊκή δράση. Αλλά τα πολιτικά κόμματα, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, η ζήτηση, τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται πολύ περισσότερο με την εθνική διάσταση. Θα έχουμε εκλογέ όπου να είναι και δυστυχώς θα έχουμε 27 ε, διαφορετικές εκλογές στις διάφορες χώρες μέλη και όχι μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Ενιά. Ακούστηκε πολλές φορές σήμερα ότι η Ευρώπη δεν προστατεύει τους πολίτες της. Αυτό είναι το κλασικό μήνυμα που μας στέλνουν οι πολίτες και που κρύβει την ουσία του προβλήματος, που είναι ότι ποιος τελικά καλείται να προστατεύσει τους πολίτες οι εθνικές κυβερνήσεις. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν ήθελε, δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τους πολίτες της από την οικονομική κρίση ή από άλλου είδους κρίσεις. Δεν έχει τα προσόντα. Ακόμα και χώρες που θεωρούνται φιλελεύθερες και που θέλουν να περιορίσουν το κράτος όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, παρόλα αυτά στις δημόσιες τους δαπάνες έχουν το 1 τρίτο του έπτους. Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ούτε καν το 1% του έπτης. Με αυτό το 1% πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύει τους πολίτες από την ανεργία, από τη φτώχεια, από ε, τα προβλήματα της νεολαίας κλπ. Δεν, μα δεν πρέπει να κορεδεύουμε τους πολίτες μας. Δεν είναι ευθύνη του ευρωπαϊκού επίπεδου να προστατεύει τους πολίτες. Αν μπορούσαμε, όπως έχει ζητήσει πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να έχουμε έναν προπολογισμό μεγαλύτερο με ίδιους πόρους, τότε θα ήμασταν σε θέση να προσφέρουμε στις χώρες μέλη αυτό το οποίο τα ίδια τα κράτη δεν μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες, την προστασία δηλαδή. Συνεπώς, θα πρέπει η σχέση των κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να γίνουν πιο στενές για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στους πολίτες ποια είναι αλήθεια. Αυτός ο διακοινοβουλευτικός διάλογος είναι πολύ σημαντικός. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε με τους επικεφαλείς των ε, κρατών και κυβερνήσεων για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά να ξέρετε ότι κανένας πρόεδρος από Εθνικό Κοινοβούλιο δεν ήρθε για να έχουμε αυτή την ίδια συζήτηση. Και σήμερα γίνεται αυτή η συνεδρίαση επειδή υπάρχει μια συγκεκριμένη έκθεση ενός ευρωβουλευτή που ζήτησε τη συζήτηση αυτή ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αλλιώς δεν θα την είχαμε αυτή τη συζήτηση. Δεν υπάρχει συνεχής διάλογος μεταξύ μας. Τέλος. Δεν λύνεται επίση το πρόβλημα με ένα κοινοβούλιο της Ευρωζώνης. Πιστεύω ότι θα δημιουργούσε περισσότερη σύγχυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρκετά δυσκολευόμαστε με ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ένα πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με μια επιτροπή, με ένα πρόεδρο της Ευρωζώνης, με ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Φτάνει αυτή η δομή. Είναι ήδη δύσκολος ο συντονισμός θα είναι πολύ πιο δύσκολο ο συντονισμό αν έχουμε και κοινοβούλιο τη Ευρωζώνη. Δεν νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δημιουργηθεί τέτοιο σώμα. Αυτό όμω που πιστεύω είναι ότι χρειάζεται ο διάλογο ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Αν δεν υπάρχει αυτός ο διάλογος, θα κυριαρχήσει η έλλειψη κατανόησης. Σε συναντώνται οι πρόεδροι του Κοινοβουλίου και στην ΑΦΚΟ πολλές φορές προτείναμε κάτι τέτοιο. Στην ιεραρχία του Κοινοβουλίου. Να κάνουμε αυτό που πρότεινες. Να ακούσουμε και τους πρόεδρους των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ποτέ όμως δεν έγινε. Δεν το δέχτηκαν. Να προσπαθήσουμε ξανά. Ευχαριστώ. Τη Δανία. Από το Forgetting Κύριος Εράσμους Νόκφιστ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Τα τελευταία χρόνια στην Δανία είχαμε διάλογο με τους πολίτες για διάφορα θέματα του ευρωπαϊκού θεματολογίου. Φέτος το έχουμε κάνει αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω της διαδικασίας διαβούλευσης με τους πολίτες. Έχουμε συνεργαστεί λοιπόν με το, την Ευρωπαϊκή Κυβέρνηση και έχουμε γυρίσει όλη τη Δανία. Δύο πράγματα έχω συγκρατήσει από το διάλογο αυτό. Όταν ρωτούσαμε τους ανθρώπους ε, ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που πρέπει να λύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είπαν οι μετανάστες ή περισσότερα χρήματα στον προπολογισμό. Όχι, ήταν το κλίμα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να συγκρατήσουμε. Κανείς δεν έχει παρουσιάσει αποτελέσματα στο θέμα αυτό. Ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε τα Εθνικά Κοινοβούλια, ούτε το Συμβούλιο, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ αυτό άκουσα επανειλημμένα από τους δανούς πολίτες. Κάτι που επίσης εμφανίστηκε πολλές φορές ήταν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι ακριβώς κάνει, πώς λειτουργεί, ποιος αποφασίζει τι. Και πολύ συχνά στη Δανία ε, λέμε ότι οι Βρυξέλλες ε, λαμβάνουν αποφάσεις, αντί να λέμε ότι ε, και εμείς συμμετέχουμε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για να λάβουμε υπόψη μας όμως στα σοβαρά το θέμα αυτό και αναφέρθηκε και, νωρί... αναφέρθηκε και νωρίτερα, τίθεται το θέμα της διαφάνειας διότι εγώ ως ε, εθνικός βουλευτής θα πρέπει να μπορώ να κάνω τη ε, δουλειά μου σωστά και να μπορώ να δω τι κάνει και το Συμβούλιο. Και δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν ε, διάφορες ομάδες εργασίας, δεν ξέρω καν τον αριθμό τους, αλλά περίπου 200 ομάδες εργασίας, όχι με πολιτικούς, που λαμβάνουν αποφάσεις και κλεισμένων των θυρών. Χρειαζόμαστε λοιπόν διαφάνεια για να μπορέσουμε να ζητήσουμε λογοδοσία από τις κυβερνήσεις μας σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνουν και να μπορούμε να εξηγήσουμε στους ψηφοφόρους μας, ώστε να μπορούν και εκείνοι να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ελήφθη η τάδε απόφαση, ε, όχι μόνο για τα κεντρικά ζητήματα, αλλά και για όλα τα άλλα. Αυτά πρόθεσμα. Περισσότερη διαφάνεια, δηλαδή. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να ε, αλλάξει μια ανοιχτή η, προ η Προεδρία. Το άλλο θέμα είναι, ωραία, πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θέλουμε να εξελίξουμε την δημοκρατία μας, πώς μπορούμε να έχουμε πολύ περισσότερο συμμετοχική δημοκρατία, ώστε να συμμετέχουν οι πολίτες και να μην λαμβάνουν μόνο οι αποφάσεις Βρυξέλλες, αλλά όλοι οι πολίτες της Ευρώπης να νιώθουν ότι αποτελούν τμήμα της Ένωσης. Ένα στοιχείο κλειδί είναι τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετέχουν ε, περισσότερο σε όλη τη διαδικασία. Αλλά επίσης ε, όταν έχουμε συναντήσεις με τους πολίτες, όταν έχουμε διάλογο με τους πολίτες και μιλάμε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, πώς μπορούν να συμμετάσχουν περισσότεροι πολίτες. Ε, σε τοπικό επίπεδο γίνονται πολλά, αλλά πώς μπορούμε να έχουμε συμμετοχική δημοκρατία στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που πρέπει να αναρωτηθούμε εάν Θέλουμε οι πολίτες να έρθουν πιο κοντά σε όλα αυτά που κάνουμε εδώ από κοινού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Από την Ιταλία, κάμερα την Τεπουτάτη. Έχουμε τον Αντρέα Κρύπτα από την Λέγκα του Βορρά. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμμετέχω σήμερα σε αυτή τη σημαντική συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης πεπισμένο ότι η κοινοβουλευτική διάσταση είναι το κλειδί για να βρούμε λύσει στα προβλήματα που είναι μπροστά στα μάτια απάντων. Με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών, που πολλέ φορέ τα τελευταία χρόνια είδαν την Ευρώπη σαν μια απόμακρη οντότητα, μακριά από του πολίτε, με κανόνε που έρχονται άνωθεν χωρί να υπάρχει αναγκαία συμμετοχή. Η Ιταλία συζητά το θέμα τη επικροπήση του εγγράφου τη νομοθεσία για τα οικονομικά δημοσιονομικά. Είναι το πρώτο έγγραφο προγραμματικό όσον αφορά τον προπολογισμό τη νέα κυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι χωρίς ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για την Ευρώπη και ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε μια ε, ερμηνεία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης μόνο από την πλευρά της λιτότητας. Είναι και η ώρα να επιδιώξουμε και το δεύτερο τμήμα του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη, δηλαδή που καλεί στην Ευρώπη να πάει προ την ε, ανάπτυξη για να παίξει ρόλο πρώτη σε έναν κόσμο που γίνεται πάντα πιο ανταγωνιστικό. Γι' αυτό το λόγο ήθελα να διαβάσω το σχέδιο ψηφίσματο, να δώσω το σχέδιο ψηφίσματο μια πιο αποφασιστική θέση επίκριση κατά των πολιτικών τη μοναδική λιτότητα που δεν οδήγησαν σε εξυγίανση των δημοσιονομικών. Η τελευταία λιγμή στην Ιταλία, οι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξηναν συνέχεια το δημόσιο χρέο, περιορίζοντα την ανάπτυξη. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα και να δώσουμε σε αυτό που ζητά αλλαγή πολιτική τουλάχιστον την αμφιβολία. Να το σκεφτούμε. Η πρόταση ψηφίσματο αναφέρεται επανειλημμένα στη λέξη ολοκλήρωση. Πρόκειται περί ενίας σημαντικής. Αλλά εμεί πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση δεν μπορεί ποτέ να σημαίνει έγκριση ή μάλλον ακύρωση τη ταυτότητά μα και των εθνικών παραδόσεων και των περιφερειακών ε, παραδόσεων που πρέπει να διατηρηθούν σαν πλούτο τη Ευρώπη. Πάνω σε αυτό ήθελα να διαβάσω πιο σαφή λόγια για την μετανάστευση, που αντιπροσωπεύει μια πτυχή κρισίμου σημασία για το μέλλον τη Ευρώπη και για το μοντέλο τη Ευρώπη που θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε κατά την άποψή μου με πεποίθηση να υποστηρίξει τα κράτη όπω είναι η Ιταλία, που θέλουν να δώσουν συγκεκριμένη συνέχεια στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που υθετήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, που ζητά από όλα τα κράτη-μέλη να κάνουν το καθήκον τους όσον αφορά την αλληλεγγύη και τον επιμερισμό του προβλήματος της μετανάστευσης. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι στο, πρόγραμμα, στο σχέδιο ψηφίσματος να γίνεται σαφής μνήα ε, ενός σταματήματος της παράνομης μετανάστευσης και ελπίζουμε τελικά τα χρήματα των Ευρωπαίων ε, φορολογωμένων να χρησιμοποιηθούν για να μην έρχονται στην, στην Ιταλία ε, κρυφά μετανάστες ε, που έρχονται από την Αφρική και είναι εις Ευρώπης. Όσον αφορά, ε, το, η, θέλω να πω ότι η Βουλή μας στην προηγούμενη θητεία, στον Φάτο το Ευρώπης, είχε εκφράσει μεγάλες απορίες όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχει έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες στη σύνθεση όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς κάποιων αποφάσεων από τον κανόνα της ομοφωνία εκείνων της ειδική πλειοψηφία. Θεωρώ ότι θα ήταν καλό να κάνουμε μια καλή αξιολόγηση των θεμάτων επί των οποίων ίσω μεγαλύτερη περιπλοκότητα ε, στι αποφάσει είναι το σωστό τίμημα για την επίτευξη μια ε, συμφωνή γνώμη και να μπορούν να συμμετέχουν και τα κράτη και οι λαοί τη Ευρώπη στι πιο μεγάλε αποφάσει. Αναφέρθηκε η ανάγκη να ενισχύσουμε το διάλογο μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίων. Με ικανοποιεί αυτή. Εμείς με πεποίθηση ακολουθήσαμε αυτό το δρόμο και ξεκίνησε, τη θητεία που ξεκίνησε, Στείλαμε έγγραφα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επί των ευρωπαϊκών θεμάτων που σημαντικά. Ευχή μα είναι μεγαλύτερη εξέταση αυτών των συνεισφορών, λαμβάνοντα υπόψη και καλύτερο συντονισμό με του ευρωβουλευτέ. Κλείνω εκφράζοντα την πεποίθηση ότι πρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλη προσοχή στο δρόμο που έχουμε, έχει ανοιχνεύσει, έχει ανοίξει η Task Force για την επικουρικότητα για να αποφύγουμε υπερβολέ ρυθμίσεων λεπτομερών από πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αφήνοντα αυτέ τι πτυχέ στα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να εγγυηθούμε καλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρουμανία. Η κυρία Γκαμπριέλα Κριτσού από την ε, γερουσία της ε, Ρουμανίας. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, εγώ ε, επί καιρών επαναλάβανα ότι μια φήμη διαδιδόταν σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή ότι η Ένωση ήδη έχει εκτελέσει το καθήκον της και μπορεί να πεθάνει πια. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την ιδέα εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η αρχή. Αντιθέτω, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την πιο ειρηνική, αναπτυγμένη και ισότιμη κοινωνία στον κόσμο. Παρά, παρά τις αυξανόμενες ανισότητες και εντάσεις. Μια Ευρώπη εθνικών κρατών μελών είναι κάτι που είχαμε πριν, στον 20ο αιώνα, και που καταλήξαμε σε δύο πολέμους Κάθε χώρα έπρεπε να ανοικοδομηθεί επί δεκαετίες μετά. Πρέπει όμως να βρούμε λύσεις σχετικά με το πώς θα διαφυλάξουμε την Ένωση, θα την κρατήσουμε ενωμένη τώρα στη δική μας γενιά και την ειρήνη, διότι η Ένωση έχει χάσει την παλιά της έγλη και γοητεία. Αυτό δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Κρατώντας ενωμένη την Ένωση μέσω φόβων κρίσεων και καμιά φορά φανταστικών κινδύνων που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η ασφαλμένη μέθοδος. Υπάρχουν πολλά πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Η Ένωση έχει πρόβλημα κατεύθυνσης. Είναι οφειλελεύθερη κατεύθυνση, για το πούμε ξεκάθαρα. Συζητούμε υπερβολικά για το πώς θα αποφασίσουμε δημοκρατικά για κάτι και σε ποιο επίπεδο πρέπει να ληφθεί η απόφαση εθνικό, ευρωπαϊκό, αλλά αυτή η προσέγγιση μας εμποδίζει από το να προσέξουμε το τι πραγματικά αποφασίζεται. Αν οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι οργισμένοι, δεν είναι λόγω των διαδικασιών λήψεων αποφάσεων. Οι πολίτες είναι στενοχωρημένοι λόγω του περιεχομένου των αποφάσεων που λαμβάνουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο εμείς και λόγω των αποτελεσμάτων που έχουν οι αποφάσεις στη ζωή τους. Στο βαθμό που η Ένωση παρέχει αποτελέσματα για όλους και αν όλοι γνώριζαν περί των αποτελεσμάτων ε, θα ήταν νόμιμη η Ένωση. Αντί να δώσουμε λύση κοινοτικό επίπεδο στην Ένωση, ποια είναι η καινούργια τάση που διαπιστώνεται. Η, η φιλοσοφία οικονομικής διακυβέρνησης λύνει προβλήματα δίνοντας ξανά στις πρωτεύουσές μας ευθύνες για κοινά προβλήματα. Αλλά δεν δουλεύει αυτή η αποκέντρωση των εξουσιών, διότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να ελέγξουν τις αγορές τους και τα νομίσματά τους. Πρέπει τα προβλήματα τα σχετικά να τα λύσουμε μαζί. Μετά, η Ένωση έχει λειτουργικό πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανεξάρτητα από πόσο ακριβή είναι, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αποτυχία των δικών μας κομμάτων το να δημιουργήσουν την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, συνομιλώντα και εισακούγοντα την άποψη των πολιτών. Η διαβούλευση στο διαδίκτυο θα μπορούσε να δημιουργήσει μια ψευδή εικόνα πραγματικότητας. Μόνο οργανωμένες ομάδες συμφερόντων έχουν δυνατότητα να καθορίσουν και να εκφράσουν τη βούλησή τους και αυτές να στέλνουν απόψεις όταν γίνεται διαβούλευση. Πέρα από τις νέες προκλήσεις, από την αρχή της Ένωσης είχαμε τρία διαθετικά προβλήματα που έπρεπε να σκεφτούμε. Κοινωνικός πυλώνας, μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η ενιαία αγορά αλλά έχουμε 27, ας πούμε 28 κοινωνικά συστήματα που υπονομεύουν τον κοινωνικό ιστό παντού. Πολύ υψηλή κινητικότητα και της αγοράς εργασίας και του κεφαλαίου και δημιουργούμε μια οικονομία χωρίς σύνορα, αλλά κοινωνίες με σύνορα. Έτσι δε περαιτέρω, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση καθιστά τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ε, ανενεργά και θα πρέπει να συνεργαστούμε για εφάνταστες νέες λύσεις, για θέσεις εργασίας που εξαφανίζονται. Έχουμε έφταστο νομισματικό σύστημα χωρίς πολιτική βούληση και ισχύ για να ολοκληρωθεί το νομισματικό σύστημα και το ευρώ να γίνει πραγματικό ενιαίο νόμισμα είναι ένα άλλο πρόβλημα. Αλλά αγαπητέ κύριε Αλμούνια, ο Υπουργό Οικονομικών χωρίς προπολογισμό που να αξίζει αυτό τον τίτλο ε, είναι μόνο κενό περιεχομένου ε, σαν λύση. Ένα κέλυφος σαν περιεχομένου. Και κλείνοντας να πω ότι εξαρτώμεθα ακόμα από τους άλλους σχετικά με την άμυνα παρά ένα πολύ υψηλό επίπεδο στατιωτικών δαπανών που γίνεται εξακολουθούμε να εξαρτώμεθα από άλλους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έλμαρ Μπροκ από το ΕΛΚ. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ θερμά και σας ευχαριστώ θερμά που μας δίνετε τη δυνατότητα να έχουμε την συζήτηση αυτή εδώ σήμερα. Ε, απλά λυπάμαι που το δικό μου Εθνικό Κοινοβούλιο δεν εκπροσωπείται εδώ σήμερα. Ίσως θα έπρεπε και εκείνοι να ε, έχουν περισσότερο ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά. Εθνικά και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί κάθε εθνικό κράτος να αντιμετωπίσει μόνο του όλες τις ε, προκλήσεις ε, που συναντά. Θα πρέπει κάποια θέματα να τα εξετάσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για παράδειγμα, νομισματική ασφάλεια. Σκεφτείτε τις κρίσεις που είχαμε. Η Ευρώπη κατάφερε ε, με πολύ επώδυνα μέτρα να αντιμετωπίσει την κρίση, κάτι που δεν θα μπορούσε να έχει γίνει σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας ότι σήμερα έχουμε κατά 19% λιγότερους ε, ε, μετανάστες από ό,τι πριν από δύο χρόνια. Στους ε, τομείς αυτούς είναι απαραίτητο να γίνονται περισσότερα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει όμως να δώσουμε και τα κατάλληλα εργαλεία στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσει από την Ευρώπη χωρίς να της δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία όταν λέμε ότι θέλουμε περισσότερο έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και το Συμβούλιο αποφασίζει ότι θα έχουμε 10.000 περισσότερους ε, συνοριοφύλακες χωρίς να προβλέψουμε τους απαραίτητους πόρους στον προϋπολογισμό, τότε δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι πρέπει να κάνει περισσότερη η Ευρώπη και να μην της δίνουμε περισσότερα χρήματα. Δεν θα λειτουργήσει αυτό. σε εθνικό επίπεδο πολύ συχνά πραγματοποιείται μια καθόλου λογική συζήτηση. Θα πρέπει να φροντίσουμε να βελτιώσουμε τους ελέγχους. Και εννοώ, το έχουμε πει αυτό επανειλημμένα, ότι χρειάζεται το Υπουργικό Συμβούλιο που υιοθετεί νομοθεσία σε αυτό το σύστημα των ε, δύο φορέων να είναι διαφανές όπως και σε ένα ομοσπονδιακό σύστημα. Είναι σημαντικό τα εθνικά κοινοβούλια να γνωρίζουν ε, ποιες ε, χώρες έχουν ψηφίσει πόσο στο Συμβούλιο. Είναι σημαντικό να το γνωρίζει αυτό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακόμα πιο σημαντικό είναι να το γνωρίζουν οι πολίτες. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσει προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν σε εθνικό επίπεδο, αλλά χωρίς να λέμε ποιος έχει ψηφίσει τι στο Συμβούλιο, ποιος αποφάσισε τι και πότε. Διότι αλλιώς δεν υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση απέναντι στους πολίτες. Και αυτό νομίζω ότι είναι αποφασιστική σημασία σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό ισχύει και για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Η νομοθεσία λοιπόν της δεύτερης βουλής, του Συμβουλίου δηλαδή, η νομοποίηση του εξαρτάται από τη διαφάνεια. Σκεφτείτε τι συμβαίνει στο Παρίσι και στο Βερολίνο. αποφασιστική σημασία παράγοντα για τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη σήμερα είναι αυτό. Και θα πρέπει να καταστεί σαφέ πού λαμβάνονται οι αποφάσει. Ο πολίτη πρέπει να γνωρίζει τι αποφασίστηκε και πού. Θα πρέπει να είναι σαφέ όμως και ποια είναι τα διάφορα επίπεδα λήψη αποφάσεων. Το χειρότερο που μπορούμε να έχουμε είναι μεικτά επίπεδα λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει να υπάρχουν σαφεί ευθύνε. Θα πρέπει να δείξουμε ότι όπου σύμφωνα με την συνθήκη έχουμε ευρωπαϊκή αρμοδιότητα θα πρέπει να αποφασίζουν τα εθνικά θεσμικά ε, όργανα, ενώ όταν έχουμε εθνική αρμοδιότητα θα πρέπει να αποφασίζουν οι εθνικοί φορείς. Τα κοινοβούλια, για παράδειγμα, και θα πρέπει να ενισχυθούν τα εθνικά κοινοβούλια, να έχουν ε, ε, ε καλύτερες ε, δυνατότητες ελέγχου ε, των κυβερνήσεών τους στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Θα πρέπει να αποτρέψουμε να ακολουθήσουμε τη λάθος κατεύθυνση Βρίσκω λοιπόν λάθος αυτήν την σύγχυση των αρμοδιοτήτων, να μην είναι σαφέ δηλαδή απέναντι στον πολίτη Ποιο φέρει την ευθύνη. Πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσουν σε αυτό. Η κίτρινη και η πορτοκαλή κάρτα και ο έλεγχος της επικουρικότητας και της αναλογικότητας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Και δεν ελέγχουμε την ορθότητα της απόφασης, ελέγχουμε το αν έχει ληφθεί στο κατάλληλο επίπεδο. Και εγώ συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και από ό,τι γνωρίζω δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής η πορτοκαλή κάρτα. Η πορτοκαλί κάρτα έχει να κάνει με την επικουρικότητα. Το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να λαμβάνουν απόφαση και να τελειώνει εκεί η νομοθετική διαδικασία χωρίς ε, η Κομισιόν να μπορεί να κάνει κάτι. Και εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να επιδιώξουμε συνέχιση αυτής της διαδικασίας. Θα πρέπει να ασχοληθούν περισσότερο με την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων και να δημιουργήσουμε και τις σχετικές διαδικασίες. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Άσο Μαλτικένια, Λιθουανία, παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου η ομιλήτρια δεν ακούγεται. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι Ευρωπαίοι πολίτες, μάλλον οι Λιθουανοί, είναι πιο αισιόδοξοι από το μέσο όρο των Ευρωπαίων για το μέλλον της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν όλο και περισσότεροι σκεπτικιστές εξαιτία κυρίως του γεγονότος ότι δεν κατανοούν πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και επειδή η ευημερία δεν είναι ισότιμα κατανεμημένη. Στη δικιά μου χώρα, οι πολιτικοί, όταν αντιλαμβάνονται ότι κάποιες αποφάσεις δεν είναι δημοφιλείς, λένε, όπως είπε πριν και ο Δανός συνάδελφος, ότι η Ευρώπη φταίει και ότι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Νύπτουν τα σχήρα τους δηλαδή. Αυτό μπορεί να ακούγεται παράδοξο, αλλά νομίζω ότι εφόσον οι χώρες διαμορφώνουν περισσότερο την πολιτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι μόνο αποδέχτες της πολιτικής, θα βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Πρέπει να σταματήσουμε την ολοκλήρωση η οποία βασίζεται σε μη ε, σε έλλειψη πραγματικότητας, απλώς σε υποθέσεις, σε εικονικές καταστάσεις τα μελλοντικά σενάρια πρέπει να βασιστούν στις χειρότερες υποθέσεις. Και στη συνέχεια για να τις αποφύγουμε, την υλοποίησή τους δηλαδή, πρέπει να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Πρέπει να υπάρχουν κοινέ κοινωνικές προδιαγραφές, να υπάρχει ένας ισχυρός κοινωνικός πυλώνας αν δεν θέλουμε τη διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. να προστατεύσουμε τις χώρες και τις περιφέρειες εφόσον χρειάζεται από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Έπειτα δεν πρέπει να υπάρξει νέα διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν δεν γίνουν οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις. Γιατί θα είναι το τελειωτικό χτύπημα αν μπουν χώρες οι οποίες δεν είναι έτοιμες και εφόσον και η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη. και μπορεί να χρειαστούν και άλλες ε, κυρώσεις αν κάποιες χώρες δεν τηρούν το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τα θέματα το μεταναστευτικό και άλλα είναι πραγματικά μεγάλα αγκάθια. Οι υποψήφιες χώρες μπορεί να απογοητευτούν Έπειτα πρέπει να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις. Η συζήτηση όμως αυτή τη φορά πρέπει να επικεντρωθεί στους πολίτες, όχι όπως έγινε την προηγούμενη φορά με την διαβούλευση για το μέλλον της Ευρώπης, γιατί πρέπει να έχουμε τη στήριξη των πολιτών. Χρειάζεται εκδημοκρατισμός των θεσμικών οργάνων και μείωση των ε, Ευρωπαίων αξιωματούχων. Όλες οι χώρες μέλη και οι νέες χώρες, η δικιά μου μεταξύ άλλων, πρέπει να αλλάξουν τη στάση τους όταν αξιολογούν την κατάσταση και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε περισσότερα, γιατί μόνο έτσι θα παίρνουμε και περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. από τις συζητήσεις αυτές θα καταλήξουμε σε κάτι που βέβαια δεν θα είναι ικανοποιητικό για όλους. Δεν είναι δυνατόν να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Αυτό είναι ουτοπία. Αλλά πρέπει να βασιστούμε στην κοινή μας νοοτροπία. Στη συζήτηση αυτή πρέπει να πούμε και τις δυσάρεστες εμπειρίες που έχουμε. Ευχαριστούμε. Πραντομπούκοβιτς Μαυροβούνη από άλλη μια υποψήφια χώρα, δηλαδή από την Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων. Έχετε το λόγο. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο. Είστε εκεί, εντάξει. Ωραία, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου, τη γλώσσα του Μαυροβουνίου. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα του ερμηνεί ε, των κρατικών που θα με βοηθήσουν να περάσω το μήνυμά μου, λέει ο μιλητής. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, σας χαιρετώ όλους και σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε και μας. Είμαστε από την Επιτροπή Στεγματικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου του Μαυροβουνίου. Ευχαριστούμε λοιπόν για την πρόσκληση. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ χρήσιμη συζήτηση αυτή που γίνεται εδώ σήμερα και για μας. Η συμμετοχή μας σε αυτό το φόρουμ, σε αυτό το βήμα, Και το αποτέλεσμα των ε, εργασιών της ε, βουλευτικής αυτής επιτροπής και της δικιάς μας Επιτροπής Δαγματικών Υποθέσεων συναντηθήκαμε στο Μαυροβούνιο και εκεί ξεκίνησαν οι απευθείες επαφές μεταξύ μας και εκεί αποφασίσαμε να έχουμε πιο συχνές συναντήσεις. Λοιπόν, εγώ προέρχομαι από μια υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι ενήμερα. Εδώ και πολύ καιρό ακούμε σχόλια που λένε ότι το Μαυροβούνιο είναι υποψήφια χώρα, ότι είμαστε μια επιτυχημένη χώρα στα Βαλκάνια και από την άλλη ακούμε ότι βρισκόμαστε σε, στην πρώτη σειρά από τις διάφορες υποένταξη χώρες. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το ότι το Μαυροβούνιο έχει επενδύσει πάρα πολύ για να ακολουθήσει το δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δρόμο της ένταξης. Δεν διστάζουμε. Είμαστε αποφασισμένοι. Όλοι αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μας ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε και εμείς τον ίδιο δρόμο. Στο στάδιο που βρισκόμαστε, που είμαστε στο δρόμο δηλαδή για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω να επαναλάβω τα λόγια του Πρόεδρου μας, ο οποίος μίλησε σε μια ειδική συνάντηση πριν από λίγο καιρό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είπε ότι χαιρόμαστε πολύ πως υποψήφια χώρα έχουμε την ευκαιρία να ενταχθούμε. Παρακολουθώ λοιπόν τη σημερινή συζήτηση και θέλω να σας μεταφέρω το εξής μήνυμα περιμένουμε ότι εν ώψη των ευρωεκλογών θα προχωρήσετε με αισιοδοξία και ότι όλα θα πάνε καλά. Τι εννοώ δηλαδή. Εννοώ ότι εύχομαι να βρεθείτε αντιμέτωποι με όσο γίνεται λιγότερα προβλήματα. Ε, προστατεύστε την Ευρωπαϊκή Ένωση σας παρακαλώ γιατί είναι η ελπίδα μας για το μέλλον. Αλλιώς όλοι εμείς, υποψήφιες χώρες και χώρες μέλη θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα ξεπεραστούμε από την ιστορία μας. Άκουσα πολύ ενδιαφέρουσες σκέψεις για μεταρρυθμίσεις εδώ. Είσαστε οι κατάλληλοι συνομιλητές μας σε αυτή τη συζήτηση. Στο Μαυροβούνιο πάντως, εμείς προστατεύουμε τις δημοκρατικές αξίες και όταν ενταχθούμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια θα είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. Αυτές τις στιγμές αστάθειας στα Βαλκάνια, το Μαυροβούνιο αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο, γιατί είμαστε Ευρωπαίοι όσον αφορά τον πολιτισμό μας, τις παραδόσεις μας, αλλά και τις πολιτικές μας θέσεις. το Μαυροβούνιο σας, σας στηρίζει. Ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ας ελπίσουμε ότι όλα τα όνειρα θα βγουν αληθινά μια μέρα. Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Βουλή των Λόρδων. Ο Λόρδος Τσάρλς Κίνολ. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Φοβάμαι ότι θα καλύψω παρόμοιες έννοιες που εύγλωτα εκαλύφθησαν από τον συνάδελφο Ρότζερ Λίτλ προλίγου. Υπάρχει ένα ρητό, νομικό, ότι ο δικαστής ακούει το επιχείρημά σου μόνο το επαναλάβει την τρίτη φορά. Και ίσως καλό θα ήταν να επαναλάβω αυτά που είπα. Θέλω να επαναλάβω δύο σημεία. Όλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο θέλουν να ευημερήσει και να προοδεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέω αυτό με κάθε πεποίθηση. Είναι προ όφελο ε, των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου. Είτε θέλουμε, όπω εγώ, μια, ένα ζωηρό ε, δημοκρατικό εγχείρημα όπω είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να νικήσει, ή αν θέλω έναν ευημερούντα ισχυρό, σταθερό γείτονα και εμπορικό εταίρο σε μια ειρηνική Ευρώπη. Αυτή η μορφή είναι εξαιρετικά σημαντική στα πλαίσια της διαδικασίας ε, αλλαγών που θα οδηγήσουν ε, στο να ευημερήσει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Όλα τα θέματα είναι επιτάπητος. Συγχαίρω θερμά εκείνους που ετοίμασαν τα έγγραφα ενημέρωσης και το σχέδιο εκθέσεως. Είναι έγγραφα που βοηθούν τη συζήτηση Υπήρξε υγιή ποικιλόμορφη απόψεων που εξεφράστηκε. Υπήρξε όμως ένα κοινό θέμα που εντοπίζει κανείς ακούγοντας κάθε ομιλητή. Ποιο είναι αυτό. Να μην υπάρξει αλλαγή δεν είναι η σοφή επιλογή. Δεύτερο, η συμμετοχή των κοινοβουλίων. Στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της Βουλής των Λόρδων ε, είμαστε αφοσιωμένοι σε αυτή την προσπάθεια. Ταξιδεύουμε πολύ. Δεχόμαστε πολλές κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες στο Λονδίνο και αυτό αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του Brexit. Και έχουμε δύο ομάδες εδώ παρούσες. Είναι ο Ρότζερ και εγώ. Και μετά ο Μάικλ Τζέι είναι επικεφαλής άλλης ομάδας που είναι παρούσα εδώ αυτή η ομάδα για άλλα ζητήματα. Και Μα αρέσουν βήματα συζητήσεων όπω είναι το παρόν και η ΚΟΖΑΚ στο μέλλον. Θα θέλαμε να προσκληθούμε, να συμμετάσχουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Διότι ω βουλευτέ ε, γειτονικών χωρών έχουμε πολλέ κοινέ ανησυχίε. Κάποιε από αυτέ αναφέρθηκαν από άλλου ομιλητέ. Έχουμε κοινή ανησυχία την ασφάλεια. Οι βουλευτέ πρέπει αυτόν το συζητήσουν. Κοινή ανησυχία τη άμυνα ενώπιον δυσχερεστά των ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Απίστευτα σημαντικό θέμα. Έχουμε κοινή ανησυχία για τα οικονομικά ζητήματα. Υπάρχει απίστευτη αλληλεξάρτηση των χρηματοπιστικών υπηρεσιών και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κοινή ανησυχία για την αλλαγή του κλίματος και πολλά, πολλά άλλα κοινά συμφέροντα και ενδιαφέροντα. Αναφερόμενος σε κοινά προβλήματα πρέπει να προωθήσει κανείς και κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για όλους τους πολίτες. Κοινή αντίληψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας διαβεβαιώ ότι σε αυτή την Επιτροπή υπάρχει ευαισθησία για όλα τα αναφερθέντα θέματα. Είναι σημαντικά για τις μελλοντικέ σχέσεις. Πιστεύω επίσης ότι μπορούμε να δεσμευτούμε σαν μέλη του Ευρωκοινοβουλίου και λυπάμαι που το λέω αυτό, ότι δεν φιδόμεθα προσπαθίας να δημιουργηθεί το ταχύτερο δυνατό αντιπροσωπή Ευρωπαϊκή Ενώσεω Ηνωμένου Βασιλείου για να συνεχιστούν οι συζητήσει και ανταλλαγέ υπόψεων, αν πραγματοποιηθεί το Brexit. Ναι, πολύ καλό, λέει ο Λόρδος. Ε, Πρόσδεκτα, ναι, σε ευχαριστώ γι' αυτό. Η γερουσία της Ρουμανίας. Ο κ. Καλάτε Τίτους. Thank <clears throat> uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης πρέπει να εξετάσουμε και τις δύο διαστάσεις. Και το εγγύς μέλλον κάτι που είναι φυσικό διότι θα αναλάβουμε την Προεδρία του Συμβουλίου την 1η Ιανουαρίου 2019. Πρέπει να εξετάσουμε όμως και το απότερο μέλλον και βλέπουμε και ευκαιρίες και προκλήσεις και θα προσπαθήσουμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας μας να εξετάσουμε και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες. Όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης όμως, θα πρέπει να τονίσουμε ότι μιλάμε για το κοινό μας μέλλον που θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για τη συζήτησή μας. Αυτό θα απαιτήσει πολιτική βούληση, όραμα, στρατηγική σκέψη και σοφία, διότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς για να καλύψουμε όλα τα συμφέροντα των κρατών μελών. Θα πρέπει επίσης να αποφύγουμε να έχουμε Νέε γραμμές διχασμού στην Ευρώπη. Και τέλο χρειάζεται ειλικρίνεια στα καθήκοντά μα και θα επανέλθω σε αυτό στο τέλος της παρέμβασή μου. Η Ρουμανική Προεδρία θα προσπαθήσει να είναι ειλικρινής διαμεσολαβητής για να χειριστούμε τα θέματα που ε, θα έχουμε στο τραπέζι μας και να εξετάσουμε την εθνική και περιφερειακή προοπτική, προερχόμαστε από την Ανατολική Ευρώπη, θα πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε και διαφόρων ειδών προκλήσεις. Καταρχάς, θα έχουμε την στιγμή του Brexit κατά τη διάρκεια της ε, προεδρίας μας και θα ήθελα εδώ να σας παραπέμψω στην παρέμβαση του Λόρδου Λίτλ. Μπορεί να μας αρέσει η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου, τη σεβόμαστε όμως. Επίσης θα έχουμε τη συζήτηση για ε, τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, την προεκλογική εκστρατεία, την ολοκλήρωση της ε, προεκλογικής εκστρατείας και την ολοκλήρωση της Προεδρίας μας τον Ιούνιο. Όσον αφορά τις εκλογές, θα πρέπει να αναφέρουμε ένα στοιχείο. σε αντίθεση με αυτό που ίσχυε ίσως μέχρι τώρα, που τα συμφέροντα των διαφόρων πολιτικών οικογενειών επικεντρώνονταν στο πόσες ψήφους είχαμε, πόσους ε, ευρωβουλευτές, ε, το ΕΛ και οι σοσιαλιστές κλπ. Νομίζω ότι αυτή τη φορά άκρας σημασίας θα είναι να έχουν ισχυρή πλειοψηφία οι φωνές υπέρ της Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω έτσι να έχουμε αλλαγή προτύπου. Δεν είμαι βέβαιος αν είμαστε έτοιμοι να σκεφτούμε υπό αυτό το φως αυτή τη στιγμή. Εμείς θα θέλαμε να προσφέρουμε για την επόμενη πενταετία 2019 με 2024 ένα όραμα για την Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος του άτυπου συμβουλίου στις 19 Μαΐου στην χώρα μου του χρόνου. με τους εταίρους μας στο τρίο των Προεδριών, την Αυστρία και την ε, Φιλανδία, θα... Έχουμε επιλέξει τις τέσσερις βασικές προτεραιότητές μας ανάπτυξη, σύγκληση, ανταγωνισμός ε, και συνοχή. Διότι συνεχίζει να είναι απαραίτητη η συνοχή για πολλά κράτη-μέλη, μεταξύ άλλων της Ανατολικής Ευρώπης. Ε, τρομοκρατία, μετανάστευση και αυτό που ανέφερε άλλος Βρετανός Ευρωβουλευτής, ε, τις ε, προκλήσεις όσον αφορά την ασφάλεια από την Ανατολική Ευρώπη. Τρίτον, η Ευρώπη ως παγκόσμιος παράγοντας και τέλος, εξίσου σημαντικό όμως, οι ευρωπαϊκές αξίες. Η κυβέρνησή μας δέχτηκε να συμπεριλάβει κατόπιν δικής μας παρότρινσης και ένα θέμα για την ε, αλληλοκατανόηση και την ε, ένταξη ε, και καταπολέμηση του ρατσισμού και της ρητορική του μίσους. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική. Όλα αυτά τα θέματα θα συμπεριληφθούν στις προτεραιότητες της Ρουμανικής Προεδρίας. Δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Αξιοπιστία της ε, ευρωπαϊκής διαδικασίας. Αναφέρθηκα σε διάφορα είδη προκλήσεων. Στι χώρες μας όμως είναι σημαντικό κατά τη συζήτηση με τους πολίτε μας να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ε, ποια είναι τα σημαντικά ευρωπαϊκά θέματα και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που οδηγούν σε ε, μειωμένη εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ένα ή δύο κράτη-μέλη, για παράδειγμα, σε μόνιμη βάση απορρίπτουν απόφαση για πρόσβαση στον τομέα Σέγγεν για δύο κράτη-μέλη που οι αρνήσεις αυτές δεν βασίζονται σε κριτήρια αλλά σε πολιτική βούληση. Αυτό οδηγεί σε δυσαρέσκεια στη δική μου χώρα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς να υποστηρίξω το αίσθημα υπέρ της Ευρώπης. Πρέπει να γίνει κατανοητός ο μηχανισμός ε, της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και ο τρόπος λήψης αποφάσεων. Και τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει να καταλάβουμε περισσότερο εις βάθος τα κράτη-μέλη και τα κράτη της γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε όλοι όμοιοι. Και πρέπει να κοιτάξουμε τις γειτονικές μας χώρες, όχι μόνο νότια, όχι μόνο τα Βαλκάνια και προς Ανατολάς. Πρέπει να κοιτάξουμε και να μην παγώσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική για κάποιες χώρες, αναφέρομαι στη Μολδαβία. Επειδή πρόκειται για πολύπλοκη υπόθεση. Και τελευταία μου παρατήρηση, μια από τις προτεραιότητες θα πρέπει να είναι να αποφύγουμε τις νέε διαιρέσει στην Ευρώπη και να είμαστε ειλικρινεί στις αξιολογήσει μα και στις αποφάσεις μας. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κόβετσικ τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα συζητάμε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα διαμορφωθεί αυτό. Εγώ πιστεύω ότι για να πετύχει ένα σχέδιο θα πρέπει να εκτιμήσουμε σωστά το τι συμβαίνει τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε. Μερικοί όμως άνθρωποι ονειρεύονται. Αν σταματήσουμε θα καταλάβουμε και ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες δεν ταυτίζονται με τον σημερινό ρυθμό ολοκλήρωσης, με την υπερβολική νομοθετική ρύθμιση. Οι πολίτες στέλνουν μηνύματα στους Ευρωπαίους πολιτικούς και μάλιστα πολλά έχουν απορρίψει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα με δημοψηφίσματα και έχουμε και το Brexit. Οπότε οποιαδήποτε πίεση για επιπλέον ευάθυση ή πολιτική ολοκλήρωση θα ενισχύσει την αντιπαράθεση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ίδια την Ευρώπη. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται βαθιές αλλαγές. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό το γεγονός. Δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει Ευρωπαϊκό Δήμο. Δεν πρέπει να βλέπουμε τις χώρες μέλη σαν το χειρότερο κακό και το μεγαλύτερο κίνδυνο για την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη πέρασε από σύγκρουση η οποία δεν έχει να κάνει με τα κράτη-έθνη, έχει να κάνει με ιδεολογίες εχθρικές προς την ελευθερία των ατόμων. Εκεί, από εκεί οφείλονται και απορρέουν οι συγκρούσεις που είχε στο παρελθόν η Ευρώπη. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες που δεν είναι αποτελεσματικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να επιστρέψουν στο εθνικό επίπεδο. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει λιγότερα, αλλά περισσότερο αποτελεσματικά. Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για τις πολιτικές και για τους τρόπους στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό η Ευρώπη θα πρέπει να υιοθετήσει την έννοια της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων. Όσες χώρες θέλουν πιο γρήγορα ολοκλήρωση να μπορούν να την πετύχουν, αλλά εκείνες οι χώρες οι οποίες δεν βλέπουν να είναι κάτι που τους ταιριάζει να μπορούν να το αποφύγουν. Χτες συμμετείχα σε μια διακοινοβουλευτική συνάντηση όπου συζητήθηκε η οικονομία. Ήταν εθνικοί βουλευτές παρόντες και ευρωβουλευτές και ακούστηκαν πολλές και διαφορετικές ιδέες για την ε, μελλοντική Ευρώπη. Υπήρχαν ε, κομμουνιστικές ιδέες από κάποιους βουλευτές Άλλοι βλέπουν την Ευρώπη σαν τον Τιτανικό που βουλιάζει. Οι ευρωβουλευτές είπαν ότι η Ευρώπη βουλιάζει από τα χρέη και πρέπει να γίνουν περικοπές. Υπάρχει λοιπόν μια πληθώρα απόψεων, συνεπώς δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό. Πρέπει πραγματικά να επιτρέψουμε στις χώρες μέλη να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να προχωρήσουν και να συνεργάζονται με τις υπόλοιπες χώρες μέλη σε όποιο βαθμό επιθυμούν. Δεν θέλω να επιβάλλω τη δικιά μου άποψη σε έναν Πορτογάλο κομμουνιστή βουλευτή για παράδειγμα. Αλλά κάτι άλλο μπορεί να μην ταιριάζει στη τσεχική δημοκρατία. Νομίζω όμως ότι θα ήταν καλό να δώσουμε περισσότερες εξουσίες στα εθνικά κοινοβούλια. Πιστεύω ότι ο ρόλος των κρατών εθνών στην ευρωπαϊκή πολιτική γίνεται πάρα πολύ λίγο. Η κάρτες, η κίτρινη κάρτα και τα λοιπά δεν χρησιμοποιούνται ή ελάχιστα. Ήταν πολύ χρήσιμο που είμαστε εδώ και ανταλλάσσουμε απόψεις, αλλά ακόμα και σε αυτήν εδώ τη συνάντηση σήμερα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε μια κοινή γραμμή. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει κάθε χώρα να μπορεί να προχωράσει την ολοκλήρωση σε όποιο βαθμό επιθυμεί και τη ταιριάζει. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων, τα οποία θα μπορούν να παίξουν το δικό τους ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό θα ήταν ένα πρώτο βήμα για να μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο παραδέχονται ακόμα και οι πιο πιστοί οπαδοί της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αν δεν παραιτηθούμε από το όνειρο της, ε, του σούπερ κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σούπερ κράτους, δεν θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να αρχίσουμε να οικοδομούμε εκ νέου την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ε, μια διακυβερνητική συνεργασία πιο πολύ. Όσοι θέλουν, έχει καλός. Αλλιώς η Ευρώπη θα χάσει εντελώς την εμπιστοσύνη των πολιτών και όλο και περισσότερο λαϊκίστικα κόμματα θα υπερισχύουν σε βάρος των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων, τόσο στις παλιές όσο και στις νέες χώρες. Αυτά τα κόμματα, τα λαϊκίστικα, ενισχύονται γιατί τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα δεν είναι ικανά να παραδεχτούν ότι το σχέδιο αυτό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει ξεπεράσει το κατάλληλο σημείο. Ευχαριστούμε Ισπανία. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας επέτρεψε να έχουμε αυτή τη συζήτηση, αυτή την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των διαφόρων χωρών. Ευχαριστούμε τον εισηγητή, τον Ραμόν Χαρμπερή, για την έκθεσή του. Και θα αρχίσω από το τελευταίο εγώ πιστεύω ότι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τους Ευρωπαίους τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 60 χρόνια, είναι ακριβώς το όνειρο. Ότι έχουμε την ικανότητα να ονειρευόμαστε, ότι θα ξεπεράσουμε τους πολέμους, ότι θα προσφέρουμε ένα κράτος ευημερία με ισχυρούς θεσμούς, με κυριαρχία που μας έκανε Ευρωπαίους πολίτες Γι' αυτό και εγώ αποφεύγω αυτές τις συζητήσεις, αυτούς τους λόγους που είναι επικρίσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκή Ένωσης και πολλές φορές, όχι πάντα, πολλές φορές πίσω από τέτοιες ομιλίες κρύβεται η αποτυχία των ε, ίδιων που εκφράζουν αυτές τις απόψεις και τα φορτώνουν όλα στην Ευρώπη. Εγώ Θέλω την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω ό,τι θετικό υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα ε, είναι αντιμέτωπη με πολλούς διεθνείς παράγοντες που δεν θέλουν τίποτα άλλο παρά την αποτυχία της. Πρέπει να ενισχύσουμε για παράδειγμα, την δημοσιονομική μας ικανότητα, να αυξήσουμε τον προπολογισμό μας για να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Να ενισχυθεί η κοινωνική μας πολιτική είναι κάτι το οποίο ζητούν οι πολίτες μας. Και πάνω απ' όλα να υιοθετούμε πολιτικές που φέρνουν πιο κοντά τον πολίτη στην Ευρώπη. Δεύτερον, κάτι που συνδέεται και με το πρώτο, οι εθνικές κυβερνήσεις δεν μπορεί να φορτώνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ευθύνη για τα πάντα. Μην ξεχνάμε ότι οι εθνικές κυβερνήσεις εκπροσωπούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετούν και εγκρίνουν αποφάσεις. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνεται για την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι άδικο οι εθνικές κυβερνήσεις πάντα να τα φορτώνουν στην Ευρώπη όπως είπαν και άλλοι προηγουμένως αντί να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και να τα λύνουν. Πριν από ένα χρόνο το Συμβούλιο Δήμων και Κοινοτήτων έκανε την ίδια συζήτηση στο Μάστριχτ. Εκεί δηλαδή συζητήσαμε πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα η προοπτική ήταν διαφορετική, έτσι το πρίσμα. Καταλήξαμε όμως σε δύο βασικά συμπεράσματα. Το πρώτο ήταν η Ευρώπη των πολιτών. Άκουσα κάτι πολύ ενδιαφέρον για μια ενισχυμένη ευρωπαϊκή κοινή γνώμη από τον ίδιο τον εισηγητή πριν. Για να πετύχει όμως αυτός ο στόχος είναι πολύ σημαντικό να βασιστούμε στις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Οι τοπικές αρχές είναι εκείνες που μπορούν να βοηθήσουν να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη και να φέρουν πιο κοντά στον πολίτη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, οι τοπικές αρχές να συμμετέχουν γιατί έτσι θα γίνει περισσότερο αισθητή η ευρωπαϊκή ταυτότητα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τέλος. Με απασχολεί πολύ η εξέλιξη. Περάσαμε από τον ευροσκεπτικισμό στην ευρωφοβία. Γιατί σήμερα πολλοί φοβούνται την Ευρώπη. Υπάρχουν διάφορα κόμματα, πρέπει να το πούμε, στην Ευρώπη, που ενισχύουν το φόβο. Και μάλιστα δεν βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, θέλουν να δημιουργήσουν αυτό το φόβο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να την καταστρέψουν εκ των έσω. Γι' αυτό μου άρεσε αυτά που είπε ο Χαβιέρα Αλμούνια. Το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτός ο φόβος με τα κοινωνικά, με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Εγώ δεν συμφωνώ με ερμηνείε που άκουσα εδώ πέρα για την μετανάστευση. Η μετανάστευση τι είναι, είναι πολίτες άλλων χωρών που φεύγουν γιατί κινδυνεύουν να πεθάνουν εκεί είτε εξαιτία του πολέμου είτε εξαιτία της πείνας. Πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη απέναντι σε αυτά τα πλάτη και τα μήκη της γης που υποφέρουν. Συντεταγμένα, συμφωνώ, με τρόπο ώστε όλοι να νιώθουν ασφάλεια μέσα στα σύνορα. Αλλά δεν συμφωνώ και δεν ταυτίζομαι καθόλου με κάποια πράγματα που άκουσα σε αυτή την αίθουσα, γιατί πιστεύω, τέλο πάντων δεν θα συνεχίσω, αλλά δεν νομίζω ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε το μεταναστευτικό. Πρέπει να είμαστε λογικοί και να αντιμετωπίζουμε το μεταναστευτικό με λογική. Πρόκειται για ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Και τελειώνω όπως ξεκίνησα. Θέλουμε περισσότερη Ευρώπη. Λύνονται τα προβλήματα της Ευρώπης με περισσότερη Ευρώπη, με περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι θέλουν να περιορίσουν, να υποβιβάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δράση της, να ξέρουν ότι αυτό θα είναι καταστροφικό για το μέλλον της Ευρώπης και για το μέλλον των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ, Σεστά, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κυρία Μαγκίνες έχει το λόγο. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις που εξεφράστησαν. Δεν ήμουν στην αίθουσα για το απόγευμα, με ενημέρωνα από το γραφείο μου για την πολύ πλούσια και ποικίλη συζήτηση. Με την κυρία Χούπνερ συναντόμαστε συχνά με εθνικούς βουλευτές και επίσημα και ανεπίσημα. Και πάντα με γιατί καμία φορά υπάρχει ένα συνέστημα ανταγωνισμού μεταξύ μας, όταν στην πράξη έχουμε εκλεγεί από τους πολίτες να κάνουν την ίδια δουλειά σε διαφορετικά θεσμικά όργανα. Και θα ελπίζα αυτό να είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε ενδελεχέστερα, διότι εσείς από τα Εθνικά Κοινοβούλια και εγώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι σύμμαχοι είμαστε εκλεγμένοι εκπρόσωποι και έχουμε ρόλο στα συγκεκριμένα θεσμικά όργανα στα οποία υπηρετούμε. Ανησυχώ πάντα όταν ακούω σχόλια του τύπου δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό που έχει νόημα. Μας υποχρεώνει ο πολιτικός κόσμος να βρούμε συμβιβασμούς συνεχώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί από αυτής της βάσεως. Δεν σημαίνει ότι είμαστε αδύναμοι αυτό. Σημαίνει ότι είμαστε πραγματιστές και βρίσκουμε λύσεις. Όταν διαφορετικά δεν θα υπήρχε ουδέμια πρόοδος. Και όπως βλέπετε βρίσκω και μια λύση με τη... όσον αφορά την αντιλιά που με τυφλώνει αντί να λιθορίζω στα σκοτεινά. Ε, πρέπει να έχουμε επίγνωση των ρόλων που έχουμε. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια σε όλα τα κράτη-μέλη και σέβομαι και εκείνους που υπηρετούν στην τοπική αυτοδίκηση. Όλοι παίζουμε σημαντικό ρόλο όσον αφορά την παρούσα μορφή και μελλοντική της Ευρώπης. Ένα από τα ωφέλη με μικρό ωμέγα, το λέω αυτό το ωφέλη, του Brexit με μεγάλο β, είναι ότι καλύτερα είμαστε καλύτεροι, καλύτερα ενήμεροι για την Ευρώπη οι πολίτες. Συζητούμε θέματα όπως τα Ελληνική Ένωση, η ενιαία αγορά, η ελεύθερη διακίνηση, η ελευθερία μετακίνησης των κατοικιδίων ζώων, αυτά που θεωρούμε ως δεδομένα, αλλά δεν θα έπρεπε να τα θεωρούμε δεδομένα, διότι συμβαίνουν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των δομών αυτής. Μιλάμε πολύ για ρύθμιση και κανονισμούς. Δεν θα μπορούσαμε χωρίς ρύθμιση να ζήσουμε. Ίσως θα έπρεπε να τα καταφέρουμε καλύτερα, αλλά ποτέ δεν θα έχουμε ανεπτυγμένη κοινωνία η οποία δεν θα έχει κάποια, κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο προς όφελος των πολιτών. Δεν δέχομαι εκείνους που λέγουν ότι απορρίπτεται τους πολίτες της Ευρώπη. Όπως και άλλοι, και εγώ σκέφτομαι γιατί συνέβη το Brexit και λυπούμε που συνέβη το Brexit και συζητούσαμε με κάποιους συναδέλφους από το δικό μου κράτος μέλους, εκπροσώπους της περιφέρειας. Και ήταν πολύ δύσκολη συζήτηση, διότι η Ιρλανδία αισθάνεται τον πόνο του Brexit σε μεγαλύτερο βάθος, λόγω του θέματος του, της νήσου της Ιρλανδίας. Και νομίζω ότι εκτιμούμε και την έννοια της αλληλεγγύη περισσότερο και την κατανοούμε καλύτερα την αλληλεγγύη, διότι μας έχουν δείξει τόσο μεγάλη αλληλεγγύη τα 26 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, στις διαπραγματεύσεις μας σαν Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντα προσπαθώ να δω τα πράγματα από την καλή όψη, τα θετικά και όχι από την αρνητική πλευρά. Και προσπαθώ να βρω λύσεις. Ελπίζω οι ευρωεκλογέ να αφορούν ευρωπαϊκά ζητήματα και ιδεώδη. Πρέπει να πω ότι σε πολλέ χώρε δεν είναι αυτά τα θέματα, είναι θέματα εσωτερική κατανάλωση. σω τώρα είναι η στιγμή τη αλλαγή λόγω του Brexit, όπου θα είναι νοπό γεγονό στη μνήμη μας και θα μπούμε το Μάιο στην προεκλογική περίοδο συζητώντας την Ευρώπη των αξιών, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την Ευρώπη, πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη την άποψη των συναδέλφων που εδώ είπαν ότι η Ευρώπη κάνει πολλά πράγματα. Ας το κουβεντιάσουμε. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να το συζητήσουμε αντί να απομακρύνονται συνάδελφοι με καθορισμένες απόψεις. Έχω ένα σύνθημα το οποίο ακολουθώ, δεν δικό μου. Είναι χρήσιμο καμιά φορά πριν αποφασίσουμε να το ανοίξουμε το πνεύμα μας και καμιά φορά το λέω και στον εαυτό μου, όπως το κάνω και σε συναδέλφους. Ο ρόλος που παίζω μαζί με την κυρία Χούμπνερ, ο ρόλος που διαδραματίζω, ελπίζω να είναι κάτι που εκτιμάτε. Ότι εκτιμούμε την παρουσία σε εδώ και ξέρω ότι χρειάζεται χρόνος, προσπάθεια να έρθετε εδώ. Και εμείς προσπαθούμε να είμαστε μαζί με τους ε, εθνικούς βουλευτές στα πλαίσια της δομής της ΚΟΖΑΚ. Είμαστε ισχυρότεροι μαζί. Είναι γεγονός ε, της ε, ζωής. Έτσι εξελίσσονται οι πολιτισμοί. Και αυτό που είναι σημαντικό αυτέ αυτές τις συναντήσεις είναι ότι έχουμε ανταπόκριση, έχουμε αντικατοπτρισμό απόψεων τα διάφορα κάτι μέλη, κοιταζόμαστε τον καθρέφτη και δεν τα βλέπουμε όλα σαν απομονωμένες απόψεις, το ένα άκρο, το άλλο άκρο, χωρίς τίποτα διάμεσα. Πολλές φορές κλείνω τα μάτια μου και σκέφτομαι. Ας πούμε αν διαλυθεί η Ευρώπη. Ο κόσμος τι μορφή θα είχε. Διότι έχουμε ηγηθεί σε πολλούς σημαντικούς τομείς. Ήρθα μια συνεδρίαση για την ισότητα, για την αλλαγή του κλίματο για τα δικαιώματα των πολιτών, όλα αυτά τα θέματα. Εκεί ηγείται η Ευρώπη και είναι ευγνώμων η χώρα μου για αυτή την ηγεσία της Ευρώπης αυτούς τους τομείς. Για το καλό των πολιτών μας και των νέων ανδρών και γυναικών που ελπίζουμε θα ψηφίσουν, πρέπει να είμαστε ισχυρότεροι όσον αφορά την ηγεσία μας, να προωθούμε το όραμά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να σταθούμε και να υποστηρίξουμε αυτά που έχουν επιτευχθεί αντί να κλαφμυρίζουμε μερικοί από εμά περί των αποτυχιών μας, διότι πάρα πολλά πράγματα λειτουργούν. Και επιτρέψτε μου να πω ότι όταν βλέπει κανείς τη δυσκολία που αντιμετωπίζει ένα κάτω μέλος που θέλει να φύγει, πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία, διότι είμαστε τόσο βαθιά ολοκληρωμένοι και γιατί λειτουργεί το σύστημα όταν είσαι ενταγμένος. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε, Πρόεδρε, να προβώ παρατηρήσει και ευχαριστώ, συνάδελφοι, που είστε μαζί μα. Ευχαριστούμε πολύ. Άλλον ένα έχουμε από την Ισπανική Γερουσία, τον κύριο Ευαρουής. Ε, ε, κύριε Ευαρουής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να έρθουμε σήμερα. Όντως πρέπει να ακούμε με τους δε. Υπάρχει μια συμφωνία στην Ισπανία όσον, Ευρωπα... όσον αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο. Το θέμα είναι πώς θα προχωρήσουμε. Θέλω να μιλήσω για τους νέους και τη σημασία που έχουν οι νέοι σήμερα και ακόμα περισσότερο μεθαύριο. Για τις διάφορες κρίσεις που συζητάμε σήμερα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την κρίση της ταυτότητας. Τι σημαίνει για τους Ευρωπαίους η ισότητα, η ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα η Ευρώπη να φροντίζει για την ειρήνη. Κατά τη γνώμη μας η κρίση έδειξε ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή δομή. Επιβλήθηκε λιτότητα που σε πολλές χώρες οδήγησε να καταστραφεί το κοινωνικό κράτος. Ένα κοινωνικό κράτος το οποίο χρησιμεύει, βοηθάει τις κοινωνίες μας, αποτελούν δίχτυα ασφάλειας, εξασφαλίζουν την αξιοπρέπεια και τα ελάχιστα αναγκαία για να μπορεί κανείς να νιώσει ότι ανήκει και ότι είναι πολίτης. Αλλά επίσης χρειάζεται και αυτή η κοινωνική συνοχή και με την λιτότητα καταστρέφεται, καταστρέφονται ζωές και καταστρέφονται οι συλλογικές μας ταυτότητες. και ακριβώς γι' αυτό προχωράνε ιδέες που μας οδηγούν μακριά από τις αρχές και τις αξίες μας. Έχουμε μια διαφθορά η οποία καταστρέφει την οικονομία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επιδεινώθηκαν οι συνθήκε ζωής πολλών εξαιτίας της λιτότητας. Δημιουργήθηκε αβεβαιότητα, φόβος και οι άνθρωποι αυτοί ταυτίζονται με την ιδέα ότι οποιοδήποτε ξένος αποτελεί απειλή. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε ποιος είναι ακριβώς που ευθύνεται για αυτή την κατάσταση, ποιος είναι αυτός που έχει συσσωρεύσει πλούτο σε βάρος άλλων. Αυτό δεν συζητιέται ποτέ. Εμείς θεωρούμε ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν σέβεται τη Χάρτα Θεμελιωδών ε, Δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε την Ευρώπη, βεβαίως. Τη χρειαζόμαστε όλοι, ναι, καμία αμφιβολία. Αλλά πρέπει να αλλάξει το μοντέλο, το πρότυπο, να ξεπεραστούν οι σημερινέ δυσκολίε. Περισσότερη κυριαρχία, λοιπόν, που να βασίζεται στη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων κυριαρχία που να μην αποκλεί κανέναν, να είναι μια κυριαρχία ε, κυρίαρχων ε, χωρών και με τη συνύπαρξη και με έναν κοινό ορίζοντα. Συνεργασία, δημοκρατία, διαφάνεια, αλληλεγγύη, κοινωνικά δικαιώματα και πολιτικά δικαιώματα. Να προχωρήσουμε και να εξυγχρονιστούμε, να αφήσουμε πίσω την παλιά ιδέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση του Μάστριχτ και να είμαστε θαραλέοι, να ανταποκριθούμε σε αυτά που ζητάει η κοινωνία που θέλει να πάνε μπροστά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να εξελιχθούν. Εμείς επαναλαμβάνουμε την θέλησή μας και την αποφασίστικο μας υπέρ ενός χώρου δημοκρατικής Ευρώπης, γιατί πιστεύουμε ότι οι μας δεν μπορούν να προχωρήσουν με την λιτότητα. Δεν πρέπει να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια, ούτε να παρετηθούμε δεν πρέπει να προχωρούν ιδέες που είναι ολοκληρωτικές ή ο λαϊκισμός. Πρέπει να φτιάξουμε μια Ευρώπη με κοινωνική δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα και οικονομική και κοινωνική και μεταξύ ανδρών και γυναικών με έναν ορίζοντα υπέρ της κοινωνίας. Πρόεδρος, ολοκληρώθηκαν ε, οι παρεμβάσεις. Φαντάζομαι ότι ο εισηγητής μας θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μου προτείνει να συνοψίσω η πρόεδρος. Σε πέντε λεπτά θα το έχω κάνει. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ όλους από τα Εθνικά Κοινοβούλια που ήρθατε. Σας ευχαριστώ για αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστώ την πρόεδρο Χούμπνερ για την εξαιρετική αυτή ιδέα που είχε να οργανωθεί αυτή η συνάντηση. Μιλήσαμε ειλικρινά όλοι. Πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν ακούσαμε κατά της Ευρώπης έτσι λόγους. Ακούσαμε για λιγότερη Ευρώπη, για πιο μινιμαλιστική Ευρώπη, αλλά όχι κατά της Ευρώπης. Και για μένα είναι θετικό αυτό. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι υπήρξαν διαφορετικές απόψεις στην αίθουσα όσον αφορά το ποια Ευρώπη θέλουμε. Ακούσαμε όμως και δυνατές ομιλίες για μια καλύτερη Ευρώπη, για μια Ευρώπη που να ξεπερνάει τα παλιά κοινωνικά προβλήματα κλπ. Ένα βασικό κεφάλαιο στη συζήτησή μας ήταν το πλαίσιο ε, συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει κάποια δυσπιστία, το είπε και η κυρία Μαγκίνες και ο συνάδελφος Γκερέρο. Είναι λες και αναλύουμε τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, λες και είμαστε δύο πολιτικά σώματα σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Είμαστε στον ίδιο δρόμο και δεν υπάρχει διπολισμός, ούτε ανταγωνιστικές απόψεις μεταξύ μας. Πρέπει να είμαστε επικοδομητικοί. Διαπιστώνω όμως τρεις σημαντικές ιδέες. Πρώτον, προσπαθούμε να έχουμε περισσότερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Δηλαδή συμμετοχή που να εκδημοκρατεί περισσότερο την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οδηγεί στα Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, οι νομοθετικές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, πρέπει να ζητούν και την συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. Ίσως όχι με την επικουρικότητα, ίσως με προτάσεις, με πρωτοβουλίες κλπ. Και τρίτον, Υπάρχει η αναγκαιότητα συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών πολύ μεγαλύτερη στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Και αυτό το τόνισαν πολύ. Και η Επιτροπή Περιφερειών, βέβαια, αλλά όχι μόνο. Η Ιρλανδία το είπε και άλλες χώρες. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό επίσης να υπογραμμίσουμε την ανησυχία που υπάρχει από πολλούς για τις συνέπειες του Brexit. Η Ιρλανδία, να μην υπάρχει ε, ενίσχυση των συνόρων, ποιες θα είναι οι σχέσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά. Το πανεκίδι εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρέπει να προχωρήσουμε επικοδομητικά για τις μελλοντικέ μας σχέσεις. Αυτή η νέα σχέση πρέπει να ενισχυθεί και πρέπει να είναι ειδική, ιδιαίτερη. Γιατί έχουμε πολλά κοινά και δεν μπορούμε όλα αυτά να τα αφήσουμε και να τα ξεχάσουμε επειδή υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Εκφράστηκε και ανησυχία για το πώς συμμεριζόμαστε τις ευθύνες και μοιραζόμαστε μάλλον τις ευθύνες για να καθησυχάσουμε τους πολίτες όσον αφορά τις ανησυχίες τους, είτε είναι μεταναστευτικό, είτε είναι οικονομικό, είτε οτιδήποτε. Δεν μπορεί να παίζουμε πινκ-πονγκ με τις κατηγορίες για το ποιος φταίει. Η αξιοπρέπεια στην εργασία, ε, μείωση των ανισοτήτων και πολλά άλλα θέματα απαιτούν επιμερισμένη ευθύνη. Δεν μπορεί να παίζουμε βρώμικο παιχνίδι χώρες μέλη και Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποιο φταίει. Τη στιγμή που τελικά είμαστε και οι μεν και οι δε υπεύθυνοι. Κλιματική αλλαγή. Η Δανία αναφέρθηκε σε αυτό. Εμένα με εξέπληξε που κατηγορείται η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα ζητήματα. Καταλαβαίνω ότι από πλευρά της Δανίας υπάρχει επικριτική διάθεση, αλλά είμαστε στην πρώτη γραμμή, αν λάβετε υπόψη σας τι συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε στην πρώτη γραμμή σε συμφωνίες για την μείωση των εκπομπών, για τις ενεργειακές πηγές, ε, λιγότερο άνθρακα κλπ. κλπ. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνω ότι για την κλιματική αλλαγή υπάρχει ανησυχία που συμμεριζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. διαφάνεια από το Συμβούλιο. Αναφέρεται στην έκθεση στο σημείο, στην παράγραφο 8, ζητάμε να αλλάξει το Συμβούλιο και να γίνει νομοθετικό σώμα ακόμα περισσότερο με διαφάνεια. Ακούσαμε επικρίσεις για τη λιτότητα, ακούσαμε για τον κοινωνικό πυλώνα, ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνική πολιτική. Όντως και εδώ είμαστε ε, σε θέματα αρμοδιότητας κάπως πιο μπερδεμένη για το πόσο είναι των χωρών μελών και πόσο εδώ. Επίσης ακούσαμε και για διευρύνσεις από το Μαυροβούνιο, από την Τουρκία. Τα ακούσαμε και για καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία από τον εκπρόσωπο της Τουρκίας και για το μέλλον ε, των διευρύσεων από το Μαυροβούνιο. Και από τη Ρουμανία ακούσαμε τα θέματα διαφορετικών ταχυτήτων. Ο Πασκάλ Ντουάν έχει ετοιμάσει μια έκθεση για την διαφοροποιημένη ολοκλήρωση ότι τελικά την αρχιτεκτονική της μελλοντικής Ευρώπης θα πρέπει να τη δημιουργήσουμε βασιζόμενοι σε ομόκεντρους κύκλους. Ε, ίσως αρχίζοντας από την Ευρωζώνη και μετά να διευρυνόμαστε σε περισσότερες χώρες και έτσι να υπάρχει μια διαφορετική σχέση και στο τέλος να καταλήξει αυτός, ε, αυτή η ομόκεντρη κύκλη ώστε έξω-έξω να περιλαμβάνουν το ερωμένο Βασίλειο, την Ελβετία. Όπως δηλαδή και η ενισχυμένη συνεργασία, έτσι και αυτό μπορεί να καταστεί αναγκαίο στο μέλλον. Τέλος, υπάρχει ένα ρεύμα πλειοψηφικό θα έλεγα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θέλει να αντιμετωπιστεί η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης έτσι. Να έχουμε μια Ευρώπη πιο αποτελεσματική, πιο ευέλικτη, αλλά καλύτερη που να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις προκλήσεις τις οποίες εσείς αναφερθήκατε. Κοιτάξτε, να προσθέσω άλλο ένα μήνυμα από τη συζήτηση. Μετά το 2008 που αντιμετωπίζαμε πολλαπλές κρίσεις και μεγαλύτερη ανησυχία μας ήταν πώς να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από την κρίση, έπρεπε να δούμε τι έπρεπε να κάνουμε. Τώρα, όπως είπε ο Αχίμ Αλμούνια, πρέπει να δούμε το περιεχόμενο των πολιτικών. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Άλλο σημαντικό στοιχείο είναι πώς Γι' αυτό, όπως είπε και η Χακίμη στην αρχή και όπως ακούσαμε και από άλλους, τίθεται το θέμα να δημιουργήσουμε δημοκρατία, εμπιστοσύνη, ε, συμμετοχή των πολιτών, επικουρικότητα, όλα αυτά τα πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τις διαδικασίες για να είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές. Αυτό ήταν ισχυρό μήνυμα που ακούσαμε. Μήνυμα που πρέπει να ακούσουμε εμείς σαν πολιτικοί ηγέτες, διότι περί αυτού πρόκειται. Έχουμε καθήκον να κατανοήσουμε καλύτερα ότι δεν μπορούμε να επιβάλλουμε, όπως λέγατε, πράγματα στους πολίτες, τις αλλαγές, ούτε στην Ευρώπη. Πρέπει να ξεκινήσουμε διάλογο. Και όταν επιστρέψουμε στις πατρίδες μας θα πρέπει να πάρουμε μαζί μας αυτό το μήνυμα. Δηλαδή το καθήκον μας είναι πραγματικά να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τους λαούς, να αναπτύξουμε ένα διάλογο, να πηγαίνουμε στις συνεδριάσεις και αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι σήμερα δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε σαν αλλαγή εκτός αν έρθει μαζί μας ο λαός. Κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει καλύτερα, να φέρει μαζί το λαό από εμά που έχουμε εκλεγεί στα κοινοβούλια. Αυτό είναι το μήνυμα που σας αφήνω. Δύο λεπτά θα ήθελα να μου δώσετε και να σας πω κάποια πράγματα. Τι γίνεται για την προετοιμασία για τις εκλογές του χρόνου. Αποφασίσαμε ήδη ημερομηνίε 23 με 26 Μαΐου. Αποφασίσαμε στο Κοινοβούλιο χωρίς με τους Βρετανούς συναδέλφους το μελλοντικό μέγεθος του Κοινοβουλίου 705 βουλευτές, ευρωβουλευτές θα ελέξουμε, θα εκλέξουμε συγγνώμη, αποφασίσαμε όσον αφορά την κατανομή περίπου των εδρών στα κράτη-μέλη. Άρα είμαστε έτοιμοι. Αλλάξαμε επίσης τον κανονισμό για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά ιδρύματα έχουμε νέο επίτροπο, την κυρία Γιούροβα, που αναφερόταν στα νέα στοιχεία που θα επισέθουν στον κανονισμό, Αλλαγέ που σχετίζονται με τον κίνδυνο που προδημιουργήθηκε από την Cambridge Analytica, τη σχετική υπόθεση, το σκάνδαλο. Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κανονισμό για να προστατεύσουμε τι ευρωεκλογέ από τυχόν παρόμοια προβλήματα, πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, χειραγώγηση των αποτελεσμάτων θα επενδύσουμε και σε αυτό. Εδώ βρισκόμαστε. Και ελπίζουμε, όπως υπόθηκε, όπως είπε η κυρία Μαγκίνες, ότι θα μας στηρίξετε. Εκτιμούμε την υποστήριξή σας. Το θέμα των ευρωεκλογών πρέπει να είναι η Ευρώπη. Πάντα έχουμε και εσωτερικά θέματα που πρέπει να συζητούμε με, τους, με το λαό στις πατρίδες μας. Ας προσπαθήσουμε να συζητήσουμε τα ζητήματα της Ευρώπης στην προεκλογική εκστρατεία. Διότι θα χρειαστεί Χρειαζόμαστε επικοδομητικό ε, κοινοβούλιο στο μέλλον. Να συσταθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα γίνουν διαπραγματεύσει για τι μελλοντικέ σχέσει μα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν μπορούμε να σπαταλήσουμε αυτό το χρόνο του χρόνου όταν θα έχουμε τελευταία ολομέλεια ε, ο 18 Απριλίου και το νέο κοινοβούλιο θα προετοιμαστεί να ξεκινήσει να εργάζεται σκληρά το Σεπτέμβριο. Θα σχηματιστεί τον Ιούλιο το κοινοβούλιο. Ε, όλοι Πρέπει να νοιαστούμε για τις καλές συνθήκες για την Ευρώπη και τη δυνατότητα να λειτουργήσει του χρόνου όταν θα περάσουμε από δύσκολη περίοδο ε, δημιουργούνται αναταραχές, διαταραχές όσον αφορά την ε, όσον αφορά τη λειτουργία και τη σύσταση των μεγάλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Εδώ ολοκληρώνουμε τις εργασίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. ο Έλμαρκ παραπονιόταν που δεν ήρθαν οι Γερμανοί, μπορούν πάντα να έρχονται. Δεν ξέρω, πάντα έρχονται. Ε, δεν ήρθαν. Μεγάλη συμμετοχή, πολύ καλή παρουσία. Είχαμε συναδέλφου από υποψήφιε χώρε επίση, από ομάδα υποψηφίων χωρών. Σα ευχαριστώ. Σαφώ ήταν καλή συζήτηση που θα είναι χρησιμότατη για την ολοκλήρωση της εκθέσεως. Η συζήτηση για το μέλλον τη Ευρώπη θα συνεχιστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ασφαλή επιστροφή στις πατρίδες σας. Γεια σας και καλό βράδυ. Καλή επιστροφή.